Chers collègues, je vous propose de prendre place. Que nous puissions commencer notre réunion. Je veux d'abord. Ναι. Εξ ονόματος όλων μας να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της Πολωνικής Προεδρίας σας προτείνω δε αμέσως τώρα να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα διαδικαστικά. Ξεκινώντας θα ήθελα και πάλι να καλωσορίσω τους Πολωνούς Υπουργούς και να προτείνω μία ανταλλαγή απόψεων μαζί τους. Κυρία μου, η κυρία Μπιενκόφσκα, θα θέλατε ο ένας μετά τον άλλο να κάνετε τις παρουσίες σας είτε ο καθένας ξεχωριστά. Μήπως θα ήταν καλύτερα δύο Ξεχωριστά. Ναι. Η κυρία Γιολάντα Φέντακ, Υπουργό Εργασία και Κοινωνική Πολιτική, ε, σα ε, συναντήσαμε ήδη στα πλαίσια ενό τριμερού διαλόγου. Είστε και πάλι καλοδεχτοί ανάμεσά μα ε, και σα παρακαλώ να μα πάρετε σύντομα τι προτεραιότητε τη Πολωνική Προεδρία. Έχετε το λόγο. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie, ponad 30 lat temu... Σας ευχαριστώ. Εδώ και 30 χρόνια και ακόμα περισσότερα ζήσαμε μια μακρά περίοδο κρίσης ε, στην Πολωνία. Γεννήθηκε το κίνημα Solidarnos και τότε ελπίσαμε σε ένα καλύτερο μέλλον αλλά ούτε και στα πιο τολμηρά ερωτά, ε, στα τολμηρά όνειρά μας δεν θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι η Πολωνία μια μέρα θα ζούσε τέτοιες στιγμές. Και γι' αυτό ακριβώ στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής ε, και τώρα ακόμα θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή βάση, μια βάση Ευρώπη ισχυρή που να δείχνει αλληλεγγύη απέναντι στους φτωχούς, τους αποκλεισμένους, μια Ευρώπη που να δείχνει αλληλεγγύη στις γενιές που την αποτελούν. Και η Πολωνική Προεδρία θα ήθελε να σας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της. που αφορούν την αλληλεγγύη ανάμεσα στις διάφορες γενιές. Και να δούμε και το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης. Να δούμε και πώς θα έχουμε μία δραστήρια Ευρώπη, μία Ευρώπη που να εργάζεται και ακόμα με εταίρους τους πολίτες και με την κεντρική διοίκηση, της μη κυβερνητική οργανώσεις, όλους που να επιδιώκουν κοινωνικούς στόχους η αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενιές ατενίζοντας το μέλλον της Ευρώπης. Εμείς σαν Προεδρία θα θέλαμε να δώσουμε μια νέα όθηση από επαγγελματικής πλευράς και τις ενέργειες που απαιτούνται καθώς και την οργάνωση για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την επαγγελματική ζωή με την ζωή την ε, καθημερινή απέναντι στις ε, τρομερές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Λοιπόν, για την συνδυασμό αυτών των δύο πτυχών, για τη συμφιλίωση επαγγελματικής με την ε, ιδιωτική ζωή και εξετάζονται τα θέματα αυτά, πώς θα συνδυαστούν, επαναλαμβάνουμε, οι δύο αυτοί ρόλοι, όλα αυτά θα εμφανιστούν ανάγλυφα άλλωστε και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στα συμπεράσματά του. Χρειάζονται καινοτόμε ενέργειες ε, για μια πραγματική πολιτική κοινωνικής ένταξης και με την επιδίωξη και την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά και ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την απασχόληση διαφόρων κατηγοριών ατόμων όπως και των ηλικιωμένων. Να δούμε και τις θετικές πτυχές αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα λάβουμε υπόψη μας όλους τους παροτριντικούς παράγοντες και όλους τους παράγοντες που αναχαιτίζουν ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά τους επαγγελματίες να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους. Θα εκτιμήσουμε από κοινού με ποιο τρόπο η κρίση αυτή επηρέασε τις αλλαγές στην αγορά εργασίας θα δούμε και τις νέες προσεγγίσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας στα πλαίσια του 2020 και τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης θα εμφανιστούν και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου συνεργασία με τους πολίτες, η εταιρική αυτή σχέση σημαίνει διάφορες μορφές συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση, στους τοπικούς φορείς, στους μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να πετύχουμε τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Θα ήθελα να τονίσω σε όλες αυτές τις προτεραιότητες ε, τον πολύ σπουδαίο ρόλο του κοινωνικού διαλόγου, των ανταλλαγών απόψεων, των συναντήσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, ε, με τα συνδικάτα αλλά και με τους εργοδότες. Και μελλοντικά μια περίοδος δύσκολη για την Ευρώπη, ένας από τους καλύτερους τρόπους επίλυσης των κοινωνικών διενέξεων είναι να καθίσει κανείς γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να προσπαθήσει να συμφιλιώσει, να συνδυάσει διάφορα στοιχεία. Και τώρα όσον αφορά τις νομοθετικές πράξεις, προβλέπει η Πολωνία την συνέχιση των εργασιών για την αναθεώρηση της οδηγίας που έχει να κάνει με τη μητρότητα. Με τη σύνταξη του κειμένου αυτού θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα 15 χρόνια που ισχύει, εφαρμόζεται αυτή η οδηγία, τα κράτη-μέλη προώθησαν με την κατάλληλη σύνταξη τη δική τους νομοθεσία που ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας με κάποιες διαφορές βέβαια. Μερικές φορές υπάρχουν και εντελώς αποκλίνουσες απόψεις. Φαίνεται ότι για μια ενδεχόμενη συμβιβαστική λύση υπάρχει αυτή η δυνατότητα με την πρόταση λύσεων που να σέβονται κατά μεγάλο μέρος την προστασία ακριβώ την μητρότητας ή γενικότερα την γονική. Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους υπουργούς να ανταλλάξουν απόψεις ε, βάσει και της πείρας που διαθέτουν ε, σε μια άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Ελπίζουμε ότι η πολιτική ζήτηση γύρω από αυτό θα επιτρέψει ένα καινούριο άνοιγμα στα πλαίσια των εργασιών για τη σύνταξη της οδηγίας για τη μητρότητα. Θα θέλουμε επίσης να ξεκινήσουμε εργασίες πάνω στο σχέδιο μιας οδηγίας που έχει να κάνει με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό που μεταβάλλει τον κανονισμό για τον συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης επιθυμούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, πάνω σε δυνατότητες εξέβρεσης συμβαστικής λύσης και ελπίζουμε συνεργασία και άλλων αντιπροσωπιών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να πετύχουμε τον εν λόγω στόχο. Ο στόχος αυτός δεν είναι πουδενή εύκολος. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας πάνω στα σχέδια οδηγίας που αφορά την είσοδο και την παραμονή πολιτών άλλων χωρών για εποχιακή εργασία στα πλαίσια μιας εσωτερικής αλλαγής ε, μετατροπής ε, σε μια επιχείρηση και προσπαθούμε να πετύχουμε διάφορες συμβαστικές λύσεις στο Συμβούλιο. Ρυθμίσεις και σχέδια περισσότερο λεπτομερή θα εξεταστούν στη συνέχεια. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να υπάρξει μια ομάδα εργασίας για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις ομάδα εργασίας για την έντεξη, για την μετανάστευση και επίσης επιθυμούμε μια μόνιμη και σταθερή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό από το ξεκίνημα των εργασιών που διεξάγονται στο σχέδιο της οδηγίας αυτής. σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες όπως ο χρόνος εργασίες, η εξοδοτήσεως και οι αλλαγές ορισμένων οδηγιών για το εργατικό δίκαιο για να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι ας πούμε σε ναυτικές δραστηριότητε και αυτά θα αναφερθούν στην παρουσίαση του σχετικού κειμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλουμε να τονίσουμε την διάθεσή μας για να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή που ασχολείται με θέματα κοινωνικής ασφάλισης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υιοθετήσουμε την καλύτερη δυνατή θέση για όσα έχουν ήδη προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, να σας πούμε ότι ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο ΣΟΠΟΤ, μια άτυπη συνάντηση στην οποία ξεκίνησε η συζήτηση για τις προτεραιότητες που θέτουμε δύο συναντήσεις για την ενεργοπολιτική, για την απασχόληση και για την επιδεικνυόμενη αλληλεγγύη ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές εργαζομένων. Θα θέλαμε σε συναντήσεις, διασκέψεις να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που θα επικεντρωθούν ακριβώς σε παρόμοια θέματα. Και στο Βρότλαφ, ε, στην Σεπτέμβριο, θα έχουμε ε, μια συνάντηση υπουργική για θέματα για τις προτεραιότητες, για κοινωνικά θέματα εκεί. Και το κύριο θέμα αυτής της συνάντησης θα είναι η κοινωνική πολιτική, οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης και συγκεκριμένα βήματα στην οικονομική αυτή δεινή συγκυρία και άλλα προβλήματα μακροπρόθεσμα που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική του 2020 να πούμε ότι πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε και με τον πρέποντα τρόπο απέναντι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό και το Σεπτέμβριο στο Βόκλαβ στην Πολωνία έχουμε σχεδιάσει τη συνάντηση αυτή. Και τον Οκτώβριο, τον προσεχή στην Κρακοβία, προτείνουμε μια ευρωπαϊκή βάση συνάντηση κατά της φτώχειας, της ανέχειας που θα ξεκινήσει έτσι και η συζήτηση για θέματα κοινωνικού αποκλεισμού για τη μάχη κατά της φτώχειας. Μην ξεχάμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα στα πλαίσια της κρίσης. Είναι οι δύο αυτές προτεραιότητες που ελπίζουμε ότι το Δεκέμβριο θα εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα και ολοκληρώνοντας να τονίσω διάφορες ε, προτεραιότητες, πρωτοβουλίες για τις ίσες ε, ευκαιρίες ανάμεσα γυναίκες και σε άνδρες απασχόλησης και το Σεπτέμβριο στη Βαρσοβία ένα συνέδριο, μια άτυπη συνάντηση για τις ίσες ευκαιρίες ανάμεσα στα δύο φύλλα και στους μηχανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν, να συμφιλιώσουν τον επαγγελματικό με τον ίδιο, την επαγγελματική με την ιδιωτική ζωή επίσης για τις δημογραφικές αλλαγές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την απασχόληση θα εξεταστούν και αυτά τα θέματα. Όλους και όλες σας κυρίες και κύριοι σας προσκαλούμε. Ορισμένοι από εσά ήδη έχουν προσκληθεί. Θα ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στην συναντήση αυτές και συνέντευξη αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Η παρέμβασή σας ήδη έχει προκαλέσει σχεδόν όλους τους παρόντες συναδέλφους και τις παρούσες συναδέλφους να ζητήσουν το λόγο. Έχουμε όμως και την κυρία Μπιέγκοφσκα που είναι υπουργό Περιφερειακής, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οπότε έχουμε και εδώ ένα σημαντικό θέμα να δούμε, ιδίως σε σχέση με την ε, με την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος σχετικά. Οπότε, ως ε, κλασικοί βουλευτές, θα δείξουμε την απαραίτητη διαλεκτικότητα και το απαραίτητο ανοιχτό πνεύμα για να προηγηθεί ο υπουργό. Κλείνω τον κατάλογο των αγορητών λοιπόν, στα σχεδόν όλοι τους άλλους σε αυτόν και στη συνέχεια θα έχετε το καθένα το λόγο για 1,5 λεπτό εκτός των συντονιστών που θα έχουν ένα τρίλεπτο. Κυρία Υπουργέ. Ε, Σας ευχαριστώ. Όπως είπατε, Πρόεδρε, στο πλαίσιο των ζητημάτων που απασχολούν το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πολωνία, ένα από τα πιο καθαριστικά είναι η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Θα προσπαθήσω λοιπόν με λίγα λόγια να σχολιάσω το ζήτημα του Ταμείου αυτού και κυρίως το μέλλον του, διότι αυτό ενδιαφέρει την Πολωνική Προεδρία. Να ευχαριστήσω καταρχά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη τη Επιτροπή σα για το ω τώρα έργο που έχετε επιτελέσει και για τη συμβολή του Κοινοβουλίου στην πολιτική συνοχή και στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η έκθεση Πίπερ πιστεύω ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα την Πολωνική Προεδρία στο να προχωρήσουν σωστά οι σχετικές εργασίες. Θα ήθελα αμέσως να δηλώσω ότι είμαι πρόθυμη να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συζητήσω όλα τα θέματα που σας ενδιαφέρουν μαζί σας. Διότι σε αυτήν την περίοδο κρίσεως, σε αυτήν την περίοδο δυσχεριών, σε μια φάση όπου είχαμε μόλις τις 29 Ιουνίου την σχετική πρόταση, βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από την άποψη της ε, μείωσης της γραφειοκρατίας, κατά πρώτον, αλλά και από πολλές άλλες απόψεις. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ε, να δούμε πώς θα προχωρήσει η έκθεση περί και θα δούμε πώ αυτό θα επηρεάσει στην εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκό Ταμείου. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην Πολωνική Προεδρία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μάλιστα, είδαμε ότι για σκοπού προβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να συγκεντρωνόμαστε στα αποτελέσματα. Πρέπει να ξεχωρίζει η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να ακολουθείτε μια διαδικασία παρόμοια με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, λόγου χάρη για την πρόοδο του Ευρωπαϊκού Κοινού, Κοινωνικού Ταμείου. Θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να υποφεληθούμε και ενό μηχανισμού ring fencing, όπω λέγεται, ώστε να επικεντρωθούμε σε κάποια βασικότερα ζητήματα. Να δούμε πώς μπορούμε να συζητήσουμε θέματα πώς τώρα έχουν απασχολήσει τα επιμέρους κράτη-μέλη και πώς ενδεχομένως να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε δραστηριότητες κινητοποίησης και των πολιτών και ενεργούς εμπλοκής στις προσπάθειές μας. Επίσης θα χρειαστεί και μια προσπάθεια επισητιστικής στήριξης των πλέον ε, φτωχών. Εάν και προβλέπεται μια παρέκκληση από το Συμβούλιο σε σχέση με όσο τώρα έχουν αποφασιστεί. Θα πρέπει πάντως να βρούμε έναν τρόπο τελείως ε, καινούριο ώστε τα κράτη-μέλη να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα και μάλιστα στις λεπτομέρειές του. Σπέρο, ελπίζω, συγγνώμη, ελπίζω όπως είπα προηγουμένως ε, και νωρίτερα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι θα έχουμε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τις διάφορες ε, πολιτικές που θα απασχολήσουν την Πολωνική Προεδρία που θεωρεί τις πλέον εύστοχες ως προς την πρόταση κανονισμού ιδίω που αφορά και τι δικέ σα αρμοδιότητε. Αυτό θα μα απασχολήσει καθόλου το εξάμεινο τη Προεδρία μα. Όλοι αναμένουν διακαώ τι ε, προτάσει αυτέ η, Ευρωπαϊκή, η Πολωνική Προεδρία, τα κράτη-μέλη. Με τι προτάσει αυτέ θα μπορέσουμε να αναλύσουμε την κατάσταση από την άποψη την οικονομική και να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει στο σύνολό του το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θέλουμε να διεξαχθεί λοιπόν μια ευρεία συζήτηση για την συνολική προσέγγιση της ανάπτυξης με αφορμή το Ταμείο αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό παράδειγμα της ε, ολοκληρωμένης ανάπτυξης είναι λόγω χάρη η ένταξη των Ρωμά. Η Ουγγρική Προεδρία έδωσε ακριβώ την έμφαση που χρειαζόταν στο θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα όπου πραγματικά η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι η μόνη που μπορεί να ε, προβάλλει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εδώ χρειάζονται πολλαπλές μέθοδοι χρηματοδότηση και θα πρέπει όσε υπάρχουν να διατηρηθούν. Διότι ακόμα και σε αυτόν τον ε, τομέα ε, μας απασχολείται πώς θα προβληθούν σωστά οι δράσεις μας. Έπειτα υπάρχουν και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020 ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, εδώ η Πολωνική Προεδρία θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το μόνο μέσο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή ώστε να επιτεθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Ευρώπης το 2020. Ένα άλλο ζήτημα αποφασιστική σημασία θα είναι ποια σημεία θα επιλεγούν με αφορμή τη στρατηγική του 2020. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις που θα θεσπιστούν για την ε, χρηματοδότηση στις επόμενες περιόδους και προκειμένου να έχουμε ψηλή αποδοτικότητα των πολιτικών μας. Η Πολωνική Προεδρία συνεχίζει να επιμένει ότι η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών πολιτικών είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το έχουμε συνεχώς κατά νου. Μας ενδιαφέρει η απλούστευση, η αποτελεσματική λειτουργία, αλλά και η χρηστή αξιοποίηση της ε, πολιτικής αυτής, προκειμένου να δοθεί ένα παράδειγμα καλής χρήσης και για τους υπόλοιπους τομείς. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, όμως η εδαφική διάσταση, η προσοχή που θα δώσουμε στις επιμέρους περιφέρειες, επαρχίες και περιοχές είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ως προτεραιότητα. Σας καλώ μάλιστα σε μια συνδιάσκεψη που θα οργανωθεί για την αντιθετική διάσταση του Κοινωνικού Ταμείου που θα γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Βαρσοβία. Ελπίζω ότι θα έχετε λάβει τα σχετικά φυλάδια που αφορούν αυτή τη διάσκεψη, αλλά και όλες τις υπόλοιπες που θα οργανώσει η Πολωνική Προεδρία. Σας καλώ λοιπόν να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή. Θα υπάρξουν και άτυπες συζητήσεις επί και ελπίζω να είστε εκεί. Ένα άλλο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι η καλή διακυβέρνηση. Το πόσο οι διοικητικέ δηλαδή αρχέ έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τι μεταρρυθμίσει. Αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα την Πολωνία ω προ την ε, αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Να κάτι το οποίο θα εμπνεύσει στο εξάμεινό μα την Προεδρία μα. Ένα άλλο θέμα ευαίσθητο. Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο νομίζουμε ότι μπορούμε να το ενισχύσουμε και να επιτελεστεί και άλλη πρόοδος. Ως τώρα έχουμε επιδιώξει να απλουστεύσουμε τη λειτουργία του Ταμείου αυτού, να μειωθούν οι διοικητικοί φραγμοί. Αυτέ είναι προσδοκίε που εξέφρασε και το Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Και μάλιστα όχι μονομερός ή από την πλευρά μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη σχετική τη ανακοίνωση. Υπάρχουν εδώ πρωτοβουλίε του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση που αφορούν λόγω χάρη την Γεωργία. Το μέλλον λοιπόν του Ταμείου αυτού είναι ένα θέμα που το θεωρούμε ευαίσθητο πρώτη σημασία. Θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για τη συζήτηση του θέματος αυτού και τα κάτι μελη να αφιερώσουν και κάποια προσπάθεια ώστε να αναλύσουν λεπτομερώς τις προτάσεις που γίνονται μέσω της σχετικής ανακοίνωσης. Ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της απαλλαγής από τη γραφειοκρατία και της καλής διασύνδεσης του Ταμείου αυτού για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και ε, το πώ θα συνδυαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σα προσκαλώ μάλιστα το Σεπτέμβριο και σε μια σχετική διάσκεψη που θα οργανωθεί στο Ντάντσεχ. Ε, για το μέλλον του Ταμείου αυτού, τη προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, θα μπορούσαμε να έχουμε πολλέ ιδέε και για το πώ θα λειτουργήσουν οι ρήτρε εξαίρεση εδώ. Η Πολωνία σκοπεύει να ασχοληθεί ιδιαίτερω με το ζήτημα αυτό. Σα καλώ λοιπόν, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, να συνεργαστείτε μαζί μα στον τομέα αυτό διότι για να γίνουν σωστά οι διαπραγματεύσει, να διεξαχθούν σωστά οι διαπραγματεύσει, χρειάζεται ενεργό συμμετοχή και από δική σα πλευρά. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας προσκαλώ όλους στι διάφορες εκδηλώσεις και διασκέψεις που θα οργανωθούν σε αυτό το εξάμενο στην Πολωνία, θυμίζοντα ότι εν είδη συμπεράσματο θα έχουμε μια δήλωση στην ε, διάσκεψη του, στη Σύνοδο του Συμβουλίου. Θα δούμε πώς θα διαμορφώσουμε το πλαίσιο για τις διάφορες συζητήσει που προανέφερα, όπως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον συσχετισμό του με τον πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως και είμαστε στη διάθεσή σα για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ, για αυτή την ε, πρόγευση του τι θα γίνει στην Προεδρία σας. Έχουν 22 συνάδελφοι ζητήσει το λόγο και θα ήθελα κάθε φορά να μου πείτε προς ποιο υπουργό θέλετε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σα Μία από τις δύο, γιατί αλλιώς θα μπερδευτούμε. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συντονιστέ. που μπορούν να απευθυνθούν βέβαια και προς τους δύο υπουργού, τις δύο υπουργούς μάλλον. Τρία λεπτά κάθε συντονιστής. Το πολύ δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το εξαντλήσετε και και με Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τις υπουργού και να σας πω ότι πραγματικά ανακουφίστηκα ακούγοντας τις παρουσιάσεις τους. Γιατί είδα ότι σημαντικά θέματα βρίσκονται σε καλά χέρια. Καταρχήν, και προς την κυρία Φετάρ και την κυρία Βιοσκόφκα έχω να πω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να μελετήσει κανείς αυτούς τους φακέλους. Ιδίως η κυρία Βιοσκόφκα για, ε, για το φάκελο για την υποστήριξη μητρότητας. Τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι δεν συμφωνούν για το θέμα αυτό. Ε, Εντάξει, χρειαζόμαστε συμβασμό, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Ίσως μια άτυπη Υπουργική Σύνοδος θα μας βοηθήσει να προσπαθήσουμε. Η οδηγία η σχετική έφτασε στα χέρια μας. Έχουμε ορίσει εισηγητές και ελπίζουμε ότι και οι δικοί σας υπερογνώμονες μαζί με τους συζητητές μας θα μπορέσουν να συνεννοηθούν για να διευκολυνθεί ο διάλογος. Με χαρά μας θα συνεργαστούμε επικοδομητικά και ελπίζουμε μέχρι τα τέλη του έτους η οδηγία αυτή απαστολή θα είναι στα χέρια μας. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Καθυστέρησα δύο-τρία λεπτά, δεν ξέρω, ίσως εξετάσατε ήδη αυτό το θέμα. Αλλά έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε το θέμα των συντάξεων στην Ουγγαρία. Η χώρα μου αυτή τη στιγμή ξεκινά πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις και περιμένουμε να έχουμε την Λευκή ρίβλο για το θέμα στα χέρια μας, προσεχώς. Θα ήταν καλό να δοθεί μια νέα ορμή και μια ισχυρή όθηση σε αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα το θέμα του πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά και γλίγορα σε περιόδους ε, κρίσης είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν φαίνεται ελλείψεις επικοινωνίας ε, σε ορισμένε χώρες, πράγμα που δυσκολεύει τα πράγματα. Τώρα προς την κυρία Μπικόσκαφ να πω ότι όσον αφορά την ε, ε, πολιτική για το κοινωνικό ταμείο είναι καλό να βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και υπάρχουν βέβαια κάποια λεπτά θέματα όπως η διανομή τροφίμων και κατά βάση έχει ήδη εγκριθεί ένα κοινοβουλευτικό έγγραφο με πλειοψηφία. Αλλά θα πρέπει να προειδοποιήσουμε γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, έχει πάντα προβλήματα. Ευχαριστώ, Σέρκα, και μετά Μαρκή. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Να καλωσορίσω τις δύο υπουργούς. Να τους ευχηθώ η Προεδρία να στεφθεί μια επιτυχία. Μιλήσατε ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η ευθύνη. Βλέπουμε την κρίση και στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο. Είναι λίγοι εκείνοι που μπορούν να κάνουν το ίδιο όπως εσείς μια προσέγγιση και στην κοινωνική πτυχή Κυρίες μου, μπορεί να είμαστε εμείς ο μεγάλος σας σύμμαχος, ίσως καλύτερους φίλους να έχετε εδώ παρά στο Συμβούλιο και με τους σαν φίλους τους σοσιαλιστές επίσης, εγώ είμαι συντονιστής τους. Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που είπατε όπως αλληλεγγύη και λοιπά, τι ωραίο που θα είναι να μεταφραστούν στην πραγματικότητα. Και εδώ στο ολόχρονο διάγραμμα είναι και σοσιαλιστικό αυτό, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στους μετανάστες. Είμαι Ισπανός, υπάρχουν πολλοί Πολωνοί στη χώρα μου και αυτή η λεγγύη στη χώρα μου θα πρέπει να επιδειχθεί και σε αυτούς που έρχονται εκεί. Εσείς που έχετε την Προεδρία έχετε τρία θέματα, την άδεια, την προσωρινή επίσης παραμονή. Εδώ βλέπουμε ότι όλα αυτά προχωρούν ε, και θα μπορούσατε τα τελευταία προβλήματα που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο να τα λύσετε. Και εδώ γίνεται μια μάχη Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να υπάρχει ίση αντιμετώπιση για να σεβαστούμε αυτόν τον κόσμο που έρχεται στην Ευρώπη και τους εργαζόμενους μας που να μην βλέπουν ε, σαν αντιπάλους αυτούς που έρχονται και να γίνονται εχθροί τους και να υποδαβλίζονται η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Έτσι. Και εδώ ε, αυτοί η εποχιακή επίσης εργαζόμενοι που αντιμετωπίζονται άνισα. Υπήρχαν πολλοί Πολωνοί παλιότερα, όπως είπα. Εδώ επίσης το θέμα της, ε, του συνδυασμού, της συμφιλίωσης του, επαγγελματικών δραστηριοτήτων με την ιδιωτική ζωή. Θα πρέπει να προσφέρονται δυνατότητες ε, και η εργασία να μην είναι εκεί που θα υποχρεώνει τους συζύγους να εργάζονται απ' έξω και οι σύζυγοι, οι γυναίκες ε, στο σπίτι. Θα πρέπει να μην ισχύει αυτή η εικόνα, να μην εφαρμόζεται. Εδώ λοιπόν ε, εύχομαι να πραγματοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις ε, και παντού να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζονται τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Σας ευχαριστώ, δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα άλλο. Η κυρία Αρκίν και η κυρία Σρέντερ στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τις δύο υπουργού και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία στο τόσο σημαντικό έργο τους τις επόμενες έξι μήνες. Καταρχήν θα ήθελα να αντιμετωπίσω, να αντιμετωπίσω ένα θέμα που θίξατε. Αναφερθήκατε στην ελληνική μεταξύ των γενναιών. Υπάρχουν διάφορε πτυχέ. Μόλι είχαμε το πράσινο βίβλο για τι ε, συντάξει και τη μεταρρύθμιση των συντάξεων. Έχετε κάποιες απόψεις πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης αναφερθήκατε στην παράταση τους ε, ενεργού σταζιδρομίας. Δεν ξέρω, έχουμε τόσο υψηλά επίπεδα ανεργίας μεταξύ των νέων. Πώς μπορείτε να το λάβετε και αυτό υπόψη και ιδίω πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε γενικά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων, γιατί θα πρέπει να δώσουμε κάποια ε, ελπίδα. Οι νέοι χρειάζονται την ελπίδα της απασχόλησης. Επίσης αναφερθήκατε σε άλλες ε, προκλήσεις. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη όσον αφορά εκείνους που φροντίζουν κάποια άλλη μέλη της οικογένειάς τους. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να υποστηρίξετε ιδίω ε, τους ε, φροντιστές αυτό στο δημόσιο τομέα για άτομα που έχουν ανάγκες. Κατόπιν αναφερθήκατε στον κοινωνικό διάλογο και αναφερθήκατε σε συμβιβασμούς. Αλλά Υπουργέ, που πολλοί διαδηλώνουν γιατί έχουν υιοθετηθεί μέτρα λιτότητας και σωστά ή άδικα, πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα μέτρα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω είναι αυτό σωστό ή λάθος. Εγώ λέω ότι αυτή είναι η ιδέα που έχουν πολλοί. Και έχουν εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λεω ειναι αυτο σωστο η λάθο. εγω λεω οτι αυτη ειναι η ιδεα που εχουν πολλοι και εχουν εντυπωση οτι η ευρωπαικη ενωση δεν ασχολειται με του πολίτε, αλλά προσπαθεί να διασώσει το τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρω, εσείς σκοπεύετε να έχετε κάποια μέτρα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, παραδείγματο χάρη οι κοινωνικέ ρήτρε τη συνθήκη Λισαβόνα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της Ευρώπης αυτό και θα θέλω να ξέρω τι πιστεύετε για τον τόσο κρίσιμο αυτό το τομέα. Και κατόπιν προς τη συνάδελφό σας αναφερθήκατε στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και είπατε ότι θα πρέπει να λυθεί και ότι είναι το θέμα πάρα πολύ λεπτό. Μήπως θα μπορέσετε να μας αναπτύξετε λίγο τις δικές σας ε, απόψεις πάνω στα πιο λεπτά αυτά θέματα. Ευχαριστώ. Τηρήσατε και πάρα πολύ το χρόνο σας. Η κυρία Σότερ και μετά η κυρία Φιγκυρέρα. Και λυπούμε που και να κάτσετε εκεί που δεν είναι η αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα το πρωί με την κυρία Βιασκόφσκα και γι' αυτό θα ήθελα να στραφώ προς την Υπουργό κυρία Φέντακ τώρα και να περιστώ σε ένα ερώτημα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε και στην κινητικότητα σε ένα κεντρικό σημείο, αλλά δεν είπατε τίποτα σχετικό όσον αφορά αυτό που ζητιώνω στη διάσκεψη των Προέδρων όσον αφορά τους ε, απεσταλμένους εργαζόμενους και τις δυσκολίες που έχουμε αυτή τη στιγμή με την ελόγω οδηγία και τις προτάσεις της σχετικής κομισιόν. Κατά πόσο ασχολείστε εσύ με αυτό το θέμα, ποια είναι η θέση της ε, Πολωνικής Προεδρίας για αυτό το θέμα. Εσείς ε, ποια θα ήταν η λύση, που θα είχατε κατά νου ούτως ώστε να έχουμε τελικά ίση μεταχείριση των εργαζομένων εκεί που εργάζονται και τον ίδιο μισθό επίσης. Και για να μπορούν να υπάρχουν, να διατηρηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκερέιντο, Ελμέρ, και μετά οι υπουργοί έχουν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, και εγώ πολύ σύντομα ήθελα να θέσω δύο σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, θέματα που ήδη εθίγησαν εδώ. Επειδή υπάρχει επιδείνωση των ε, κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα λεγόμενα πακέτα διάσωσης με πολύ αυστηρά μέτρα λιτότητας για εργαζομένους και πληθυσμούς που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και έχουν μεγάλες ελλείψεις στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία. Όλα αυτά υποβαθμίζουν την κοινωνική δυσκολία των ε, πληθυσμών αυτών. Υπάρχει περισσότερη ανεργία και περισσότερη φτώχεια. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Η Προεδρία της Πολωνίας τι σκοπεύει να κάνει ώστε να αναλυθεί δράση και για αυτά τα προβλήματα και οικονομική και κοινωνική συνοχή αλλά και αλληλεγγύη να μην παραμείνουν μόνον εκφράσεις ή λόγια χωρίς νόημα, να υπάρξει και ένα περιεχόμενο. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι για να πω ότι ένα από τα μέσα ώστε καλύτερα να καταπολεμήσουμε την εξάπλωση της φτώχειας είναι να προβλεφθεί και ένας ελάχιστος μισθός σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρσι με το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας εγκρίναμε σχετικά μια έκθεση. Ρωτώ λοιπόν την Προεδρία της Πολωνίας εάν έχει σκοπό στην διάσκεψη του Οκτωβρίου που θα οργανωθεί να συζητήσει και το θέμα αυτό. Θα αναλάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία για τον σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Έλμερτ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ ιδιαίτερως. Ο κύριος Ζάρντονοκ, ε, ο συντονιστής μας, δεν είναι μαζί μας εδώ, δεν μπορούσε να παραβρεθεί, οπότε θα μιλήσω στη θέση του. Να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την παρουσίασή της την κυρία Φέντακ, διότι η Πολωνία 20 χρόνια μετά την αλληλεγγύη της Πολωνίας βρίσκεται πλέον σε μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει δυστυχώς την ε, μεγαλύτερη οικονομική της κρίση από όσο μπορεί κανείς να θυμηθεί. Και υπ' αυτές τις συνθήκες αυτό που εσείς μας λέτε είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Μήπως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη είναι αυτή που προκάλεσε αυτό το χάος. Μήπω η Ευρώπη ακριβώ είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Μήπω η περισσότερη Ευρώπη κάνει τα πράγματα χειρότερα από ό,τι καλύτερα. Εσείς λέτε ότι χρειάζεται αλληλεγγύη μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Νομίζω αυτό που εννοείται είναι περισσότερο αναδιαναμετικό σύστημα, ειδικά των φόρων. Περισσότερη ισορροπία λέτε μεταξύ των ε, εργαζομένων γενεών. Ε, βλέπετε όμως ότι οι εργατικές ρυθμίσεις ε, δημιουργούν προβλήματα, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, αυξάνουν την ανεργία και στρέφουν αυτούς που έχουν ήδη εργασία κατά τον αναζητούντων εργασία. Θα γίνουμε ε, επιτροπή ανεργία σε λίγο αντί για απασχόληση. Και λέτε και για τις ε, εταιρικέ σχέσεις με τους ε, πολίτες και την κοινωνία των πολιτών. Αυτή η σχέση στην Ιρλανδία κινδυνεύει να γίνει απαγορευμένη. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε πολλά αντιπαραγωγικά σεμινάρια να εργανώνονται, όπως οι διασκέψεις που αναφέρατε, αλλά οι Αμερικανοί μας έμαθαν ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε το γρασίδι να μεγαλώνει μόνο του, αλλά πρέπει να απαλλάξουμε το έδαφος και το χώμα από τα, τις πέτρες και τα χαλίκια για να μεγαλώσει το γρασίδι. Μήπω λοιπόν αντί για περισσότερε ρυθμίσει και κανονισμού χρειάζεται απλώ να βγάλουμε από το δρόμο αυτά τα εμπόδια και να αφήσουμε την αγορά, να αφήσουμε τι επιχειρήσει να προχωρήσουν, ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη και εύρωστη οικονομία. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο Παρακαλώ σύντομα όμως. Έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που επιθυμούν να σας απευθύνουν ερωτήσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και να απαντάτε σας παρακαλώ συγκεκριμένα και εσείς χωρίς γενικής φύσεως σχόλια γιατί θα έχουμε άλλες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της πολεμικής προεδρίας για να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Έχετε το λόγο κυρία μου. Θα ξεκινήσω απαντώντας στο τελευταίο ερώτημα. Σχετικά με την αλληλεγγύη και εάν μήπως η Ευρώπη είναι το πραγματικό πρόβλημα. 7% η ανάπτυξη στην Πολωνία πριν από δύο χρόνια και η ανεργία τότε ήταν στο χαμηλότερο σημείο εδώ και 20 χρόνια και άλλαξε η ηλικία συνταξιοδότησης, είχαμε νέους απασχολούμενους ακόμα και περιθωριακά άτομα βρήκαν δουλειά και κόσμος που ήταν 50-55 ετών επίσης και τώρα αντιμετωπίζουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που θα χάσουν τη δουλειά τους πολύ και όχι από φτεξιμό τους πολλοί θα κλείσουν τις επιχειρήσεις τους ε, και οι οικογένειές τους θα μείνουν στο δρόμο. Όλα αυτά αφορούν τους τα πιο ευαίσθητους, εύθραυστους, ε, τους νέους, τους ασθενείς, ε, εκείνους με προβλήματα μπροστά σε μια παρόμοια απειλή, δεν θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε την αλληλεγγύη ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους και ανάμεσα στους υπόλοιπους, αλλά να ενεργούμε με κατάλληλο τρόπο, να δούμε και τη συνεργασία ανάμεσα στις γενιές και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένω. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση στη συνδιάσκεψη που προετοιμάζουμε για το Σεπτέμβριο που μας έρχεται και αυτά τα ερωτήματα θα τεθούν και στους Υπουργούς Κοινωνικής Πολιτικής και Εργασίας. Σε όλου αυτού τους θα πρέπει να κρατήσει κανείς να εφαρμόσει την χρυσή και όσον αφορά την, ε, τα μέτρα για τη μητρότητα, το πρώτο ερώτημα το οποίο ακούσαμε, καταλαβαίνουμε ότι στον τομέα αυτό απαιτείται υποστήριξη στις μητέρες. Έτσι θα μπορέσουν να συνδυάσουν τις ε, υποχρεώσεις τους σαν μητέρες με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτό το θέμα έχει τρομερή σημασία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την αλλαγή αυτής της οδηγίας. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι το να πετύχει κανείς μια συμβιβαστική λύση θα είναι έργο ιδιαίτερα δύσκολο. Θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους όλων των ενδιαφέρων μερών. Θέλουμε, όπως είπα για παραδείγμα, να το συζητήσουμε αυτό κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης των Υπουργών για να ξεκινήσουμε κάτι το νέο, να έχουμε το κατάλληλο άνοιγμα για να προχωρήσουμε και για να μπορέσουμε να ε, έχουμε τις καλύτερες δυνατές αλλαγές. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως είναι ένα έργο ιδιαίτερα δύσκολο. Και τώρα το πρόβλημα των συντάξεων, των συνταξιοδοτήσεων και της Λευκής Βίβλου που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας προβλέπεται να δημοσιευθεί. Πριν, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας, εμείς είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό των συντάξεων κατά τη διάρκεια της συζήτησης και κατά τη σύνταξη της Λευκής Βίβλου συμμετείχαμε σε κάθε συνάντηση που οργανώθηκε πάνω στο θέμα αυτό και εκφράσαμε τη διάθεσή μας να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και μετά από την παρουσίαση της Λευκής Βίβλου. Συμφωνούμε με κάθε παρατήρηση που ακούσαμε και ότι θα πρέπει να είναι αφενός σταθερές οι συντάξεις, αλλά άλλη μεριά και οι κατάλληλες. Κατανοούμε το πρόβλημα αυτό όσον αφορά την ε, ισορροπία στα ταμεία συνταξιοδότησης αλλά και επίσης ε, τις υπερβολικές δαπάνες. Ε, αυτό, σε αυτό αναφερθήκατε και αυτό προσπάθησε να πετύχει η Ουγγαρία. Εάν είναι έτοιμη η Επιτροπή με τη λευκή της βίβλο και αν μας πούν ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο, τότε θα ασχοληθούμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και συνεχίζουμε άλλωστε τη συζήτηση και την εξέταση των θεμάτων αυτών, ιδιαίτερα σε βάθος και σε εθνικό επίπεδο. Και στις συναντήσεις αυτές, αυτές πρόκειται για ίσες ευκαιρίες για την απασχόληση επίσης. Θα ασχοληθούμε με τις ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες στην αγορά εργασία. Και αυτό θα έχει να κάνει όχι μόνο με το συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή, αλλά και για την ίση αμοιβή για ίση εργασία και για τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ίδιες για όλους, όλα αυτά θα αποτελέσουν σημείο εξέτασης από μας. Είναι βασικό σημείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε να κάνουμε και με το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και όπως και την ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων. Είναι δύσκολο βέβαια να έχουμε μια κοινή θέση για να μεταβάλουμε, να αλλάξουμε την οδηγία για την ε, κατεξοδότηση εργασία, ανατιθέμενη εργασία. Και θα συνεχίσουμε πάντως την λεπτομερή εξέταση αυτής της εργασίας διοικητικής φύσεως και περιμένουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσουμε τη θέση της για να μπούμε σε λεπτομέρειες σε αυτή την διοικητική εργασία. αν το καταφέρουμε θα βελτιώσουμε τις συνθήκες των εργαζομένων κάτω από τις οποίες εργάζονται στην αγορά εργασίας. Θα αναλάβουμε πάντως ε, την πρωτοβουλία και εμείς και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για την υποστήριξή σας και για τα ε, καλά σας λόγια όσον αφορά την πρωτοβουλία που προωθούμε για την αλληλεγγύη ανάμεσα σε διαφορετικές γένειες όπως επίσης και για την ελεγγύη απέναντι σε φτωχότερα άτομα και με τα κράτη-μέλη, με τα ευρωπαϊκά όργανα καταβάλουμε προσπάθεια για να πετύχουμε τους κοινωνικούς μας στόχους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κοινοτική πρωτοβουλία του 2020. Και υποστηρίζομαι κάθε πρωτοποριακή προσπάθεια και τη μάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και το πλαίσιο για τη συνοχή αυτή την κοινωνική και τη γεωγραφική. Και στα πλαίσια αυτής της πλατφόρμας για τη φτώχεια ε, θα σας ε, αναφέρουμε κάθε φορά τις πρόοδους που σημειώνονται, που επιτελούνται ακριβώς αυτά όλα αυτά που επιτυχώνονται στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 και επίσης για να υπάρχει μια συνεχής παρότριση για την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, σας προτείνουμε δύο σημαντικά τα οποία θα έχουμε φθηνό πρώτο επόμενο. Είσαστε όλοι σας προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, κάτι στην Πολωνία που γίνεται εδώ και τρία χρόνια. Η διάσκεψη των γυναικών για τον κοινωνικό και επαγγελματικό τους ρόλο και τις πολιτικές τους δραστηριότητες. Θα είναι σημαντικό φέτος γεγονός με ευρωπαϊκή διάσταση και επίσης θα εξετάσουμε και τα προβλήμα ίσης αντιμετώπισης ίσων ευκαιριών στα πλαίσια της μη διάκρισης στην αγορά εργασίας και στα πλαίσια της ίσης αμοιβή για την αυτή εργασία. Και τα θέματα, το θέμα της Λευκής Βίβλου νομίζω ότι δόθηκε η διαπάντηση και την αλληλεγγύη απέναντι στους νέους και πώς θα βοηθήσουμε άτομα που αναλαμβάνουν οικογένειες ε, και το πώς θα υπάρξει μια κοινωνική αρρωγή σύμφωνα και με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά και θα θέλουμε να τονίσουμε την δεύτερη ε, δραστηριότητα, πρωτοβουλία, την ενεργό Ευρώπη και σε μερικές περιοχές δεν υπάρχει δυνατότητα εξέβρεση εργασία. Άρα λοιπόν προσπάθειες για την ένταξη ατόμων που έχουν προβλήματα, είναι κάπως το περιθώριο στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά τα προβλήματα θα μας απασχολήσουν και μας στα συμβούλια και στις υπουργικές συναντήσεις γενικότερα. Και ακόμη για το θέμα της αμοιβή των μισθών που να είναι προσαρμοσμένη στην εργασία και στις ανάγκες. Θα έχουμε μια συνάντηση για το θέμα αυτό και για τις τάσεις που εμφανίζονται σε επίπεδο κρατών μελών και να υπενθυμίσουμε ότι κυρίως το επίπεδο ε, το ύψος του μισθού της αμοιβή ε, εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Είναι δική τους αρμοδιότητας. Εμείς στην Πολωνία πάντως αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία ώστε οι μισθοί και μάλιστα οι ελάχιστοι μισθοί να αποτελούν ε, αντικείμενο εξέτασης, συζήτησης και απόφασης από την τους εταίρους σε τριμερή βάση και με μια απόφαση μετά από ε, αρκετά χρόνια, τα δέκα τελευταία χρόνια η μοναδική συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με τους ελάχιστους μισθούς. Αλλά από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι όταν πρόκειται να λυθεί ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί ποτέ, παρασχάρη αυτό, πώς να διατηρηθεί η απασχόληση και πώς να εξασφαλίσουμε την ε, οικονομική ανάπτυξη, τι θα μπορούσε να γίνει. Πρώτα απ' όλα, μια από τις λύσεις θα ήταν μια κοινή συζήτηση. Στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ το προτείνουμε ώστε οι Υπουργοί Οικονομικών, οι Υπουργοί οι οποίοι υιοθετούν την ε, στατική 2020 να θετήσουν τις κατάλληλες για την αγορά εργασίας και είναι πάρα πολύ σημαντικά πώς θα μπορέσει κανείς να προχωρήσει σε εξοικονόμηση κονδυλίων και από την άλλη μεριά να διατηρηθεί μια θετική συγκυρία στην Ευρώπη και ικανοποιητικό επίπεδο απασχόλησης. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα αυτά που θα έπρεπε. Ναι, πρόεδρος, ειλικρινά Παρακαλώ, σύντομα, σύντομα, διαφορετικά δεν θα ακούσετε τις ε, ερωτήσεις των συνέλεφων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την ερώτηση της κυρίας Χάρκιν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Προέκυψαν τελείως ε, νέα θέματα και ζητήματα μετά από την ε, ε, σχετική ανακοίνωση. Μα απασχόλησε λοιπόν το πώ θα καλύψουμε τι ανάγκε των πιο φτωχών και επίση το κατά πόσον το ταμείο αυτό θα αφορά πλέον και τι γεωργικέ δραστηριότητε. Μιλώ για καινούργια θέματα βέβαια. Σε τέτοιο βαθμό που μα υποχρεώνουν να συζητήσουμε ξανά με τα κράτη-μέλη ώστε να δούμε ποια είναι τα πιο σκόπιμα μέτρα. Όλα τα κράτη μπορούν βεβαίως να μελετήσουν ε, παρκώς τα θέματα αυτά αφού λάβουν την πρόταση κανονισμού. Για την ώρα δεν έχουμε αρκετές λεπτομέρειες. Μεταξύ λοιπόν των αρμοδιοτήτων μας και αφού υποβληθεί η πρόταση κανονισμού θα φροντίσουμε να έχουμε λεπτομερέστατα ερωτηματολόγια ώστε οι αρχές της ανακοίνωσης και εφόσον εγκριθούν να μας εμπνεύσουν και να οδηγηθούμε σε έγκριση το 2014. Ευχαριστώ, αλλά για να οργανωθούμε σωστά, παρακαλώ να λέτε για ποιον είναι το ερώτημά σας πριν να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ, για ποιον είναι η ερώτησή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην κυρία Μπιέγκοφσκα ήθελα να θέσω ερώτηση, ώστε να υπάρξει και καλύτερη ισορροπία. Μπορώ. Ε, εγώ έχω ρώτηση για την κυρία Φέντακ. Συγκεκριμένα για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για το θέμα αυτό. Αυτό θα επιδιώξετε. Διότι προφανώς ε, για τα επίπεδα επιτρεπόμενης χρήσης έχουμε αλλάξει ε, τα ποσά, οπότε θα, μπορούσατε, θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία. Επίσης για τους ε, γυριότερου, είπατε ότι θα υπάρξει κάποια μέρημνα. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει το σκοπό να γίνει με, την, ε, με κάποιες ε, συμπεριφορές καταχρηστικές και επίσης για την οδηγία της διακριτικής μεταχείρισης. Τι θα γίνει με το Συμβούλιο Κοιτάξτε, αν θέσετε τρία ερωτήματα δεν πρόκειται ποτέ να λάβετε απάντηση. Α είμαστε λογικοί. Ε, τι να κάνω κι εγώ. Εάν έχετε 1,5 λεπτό και θέτετε πέντε ερωτήματα δεν πρέπει να πάρετε απάντηση. Παρακαλώ συμπτύξτε τα. Εντάξει, θα συνεχίσω όμω το 1,5 λεπτό μου. Λοιπόν, για τον ελάχιστο μισθό, φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να οριστεί σε επίπεδο κάτω μέλους. Ένα ελάχιστο εισόδημα πιστεύετε λοιπόν θα πρέπει να οριστεί σε, κράτος, σε επίπεδο κράτους μέλους για να αναλυθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. Ενάμιση λεπτό και μία ερώτηση για τον κύριο Κοζάκη. Για ποιον είναι η ερώτησή σας. ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μπορώ να την ρωτήσω. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συγκεκριμένο, πολύ ερώτημα. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι η Πολωνική Προεδρία με χαρά διαπιστώνω ότι θέλει να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Το μέσο αυτό, το κοινωνικό ταμείο μα, ε, δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να δημιουργήσουμε ίσε ευκαιρίε στην Ευρώπη. Εγώ ο ίδιος ζω με μια ειδική ανάγκη στην καθημερινότητά μου. Πρέπει λοιπόν να πω ότι περίπου το τέσσερα 100 μόνο το ποσό που προβλεπόταν έχει δαπανηθεί για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Πώ θα μπορούσε λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτή η ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια τη Πολωνική Προεδρία. Κοιτάξτε, παρακαλώ να μου λέτε σε ποια να απευθύνεστε τις δύο υπουργού, στην κυρία Φέντα και στην κυρία Μπιεύσκοβα. Δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις αλλιώ. Κυρία Κούντς. Για ποιον είναι η ερώτησή σας. Θα σα δώσω μετά το λόγο. Κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η, κυρία, η ερώτηση μου είναι για την κυρία Φεντάκ. Ως εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια μετρότητας, έχω σχετικές προσδοκίες καλές μάλιστα, από την, θετικές από την ε, Πολωνική Προεδρία. Ήδη συναντηθήκαμε με τον αρμόδιο υπουργό σα και με την Επιτροπή Ρέντινγκ και η Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων θα υποβάλει πρόταση, μάλλον προφορική ερώτηση, στην συζήτηση της Ολομέλειας όταν φτάσει εκεί το συγκεκριμένο ζήτημα, ακριβώς επειδή το Συμβούλιο το απέμπλεξε το συγκεκριμένο ντοσχέ. και μάλιστα συνέκλεινε με την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς θα μπορούσαμε από κοινού ως Κοινοβούλιο με την Πολωνική Προεδρία να επιδιώξουμε την απαραίτητη συνένεση. Ήδη έχω πει ότι με τη ρήτρα Πασερέλ, με, την, ε, με τις διάφορες οροφές που προτείνονται, με τη σταδιακή υλοποίηση των μέτρων που προτείνει το Κοινοβούλιο, μπορούμε με όλα αυτά τα στοιχεία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία παρά τις δυσχερείς συνθήκες τις οποίες όλοι διανύουμε. Τι ελπίζει λοιπόν ως προς αυτή την, ε, αυτό το στόχο η Πολωνική Προεδρία από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστούμε ο κύριος Μάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Φελάκ, είπατε ότι μια από τις προτεραιότητες σας είναι να προωθήσει την απασχόληση των ηλικιωμένων. Είχα εγώ την ευκαιρία να προετοιμάσω μία έκθεση για την δικαιοσύνη μεταξύ των Ιουνιών που είχε σαν ε, αντικείμενο το ότι το 2012 θα έχουμε το έτος του ενεργής γύρανσης. Εγώ θα ήθελα να ξέρω στην Πολωνία πώς ε, πετυχάνεται να απασχοληθούν οι ηλικιωμένοι, πώς το πετυχαίνεται, όχι με ποσοστώσει, αλλά δίνοντα ένα πραγματικό έργο. Πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε εκείνου που έχουν τόση εμπειρία. Όχι να έχουμε αντιμέτωπους τους νέους προ τους γυρότερου, όχι. Να μπορούν όλοι να συμμετάσχουν, εφόσον έχουν βέβαια την υγεία τους. Και δεύτερο θέμα, κοινωνικός διάλογος. Στη χώρα του Σεντανόρσκο πολλά μπορεί να ζητήσει κανένα. Αν μπορείτε λοιπόν να εξηγήσετε στι άλλε χώρε μέλη ποια μορφή μπορεί να έχει ένα τέτοιο κοινωνικό διάλογο, Είπατε ότι μπορούμε να έχουμε έναν διάλογο χωρί να κατεβούμε σε διαδηλώσει, με διαπραγματεύσει, με ισχυρέ οργανώσει εργαζομένων και εργοδοτών. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε πολλά να μάθουμε από την Πολωνία. Τελευταία αναλύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εσείς ε, αναφερθήκατε για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής ε, από πλευράς των αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά είναι και συχνά ο ρόλος των ε, κοινωνικών εταίρων. Ποια είναι η άποψή σας για τη σημασία του ρόλου των ε, κοινωνικών εταίρων. Σε ευχαριστούμε. Πολύ σύντομο. Στίβεν Χιούς. Ευχαριστώ προς την Υπουργό ε, Φέρακ. Δεν θα ρωτήσω κάτι για τους ε, εργαζομένους στα ταχυδρομεία. Δεν ξέρω κατά πόσον η οδηγία όταν εφαρμοστεί θα λύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί γιατί εγώ δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Ξέρετε ότι στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια εταιρεία η οποία είναι, έχει πια μια υπερβολία από την EDF ε που είναι οργανωμένη στην Ιρλανδία, έχει καταγραφεί στην Κύπρο και απασχολεί εργαζόμενους από την Πολωνία, την και διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να τη χάνουν τις ίδιες μεταχείριση όμως. Δεν ξέρω αν και εσείς καταλήγετε στο ίδιο συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε και θα σας παρακαλέσω να είσαστε κατά το δυνατόν σύντομοι. Με συγχωρείτε που παίζω το χωροφύλακα εδώ, αλλά αυτό είναι ο ρόλος μου. Ναι, σχετικά με το ερώτημα που έχει να κάνει με το τι προσδοκούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μητρότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είχαμε πει στην αρχή ότι αντιλαμβανόμαστε το ότι οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις έχουν και εντελώς αποκλίνουσες θέσεις και είναι πολύ σημαντικό να ξεφύγει κανείς από αυτό το αδιέξοδο. Θεωρούμε ότι για το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να εξευρεθεί μια λύση για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα εργαστούμε με, τις σχετικές, με σχετικές τροπολογίες σε αυτήν την οδηγία. Και με αυτές διαπραγματεύσεις θα δούμε ακριβώς, θα συνοηθούμε με όλους τους συμμετέχοντες για να πετύχουμε ένα συμβαστικό κείμενο το οποίο θα δεχτούν όλοι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι από τότε που εφαρμόζεται η κοινωνική πολιτική τα κράτη-μέλη έχουν ασκήσει την ίδια κοινωνική πολιτική αλλά με διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο τώρα σε αυτή τη φάση να εναρμονίσουμε τις προσεγγίσεις. Τουλάχιστον όμως εμείς θα καταβάλουμε μια προσπάθεια. Έχουμε καλέσει όλους τους υπουργούς να ανταλλάξουν απόψεις, θέσεις, καλές πρακτικές κλπ. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με μια καλή σωστή βάση. Θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή συμβαστική λύση αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξουν μια κάποια ευκαινησία και ευκαμψία τουλάχιστον μετά από αυτές ε, τις ε, συζητήσεις εδώ με τους υπουργούς θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτή τη συμβαστική λύση και ελπίζουμε σε μια σωστή καρποφόρα συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε ακριβώς να πετύχουμε αυτό το συμβασμό όπως είπαμε. Πολύ καλά γνωρίζω την περίπτωση αυτή που αναφέρθηκε για τους ε, παράνομα εργαζόμενους ε, ε, μέσα στην κοινωνία εργαζόμενους που εργάστηκαν και στη Γαλλία αλλά και σε άλλες βέβαια χώρες και να σας πω ότι πρέπει κανείς να καταλάβει ότι υπάρχουν εργοδότες που θέλουν να μειώσουν το, κόστο τους, το κόστος τους και αυτό για να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε τους εργαζόμενους. Αυτοί θα πρέπει να προστατευθούν ότι εργάζονται κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες ανεξάρτητα με τη χώρα στην οποία εργάζονται. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να επιτεθούμε κατά μέτωπα στο πρόβλημα αυτό στα πλαίσια ενός διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Η συμφωνία μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην εξέβρεση μιας λύσης ε, και εάν εκείνοι αυτά τα δύο μέρη μπορέσουν μεταξύ τους να βρουν μία λύση που να είναι αποδεκτή και από τα δύο ακριβώ μέρη, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για να πετύχουμε βελτιώσεις στον τομέα αυτό. Μετά είχαμε και την ερώτηση για την διακρίσεις απέναντι σε ηλικιωμένα άτομα. Στο Βρόθλαφ ε, τον φθινόπορο θα οργανώσουμε μια υπουργική συνάντηση για τις προτεραιότητες της Προεδρίας σε θέματα απασχόλησης. Θα ασχοληθούμε με τις δημογραφικές αλλαγές, ίσες ευκαιρίες για την αναζήτηση στην αναζήτηση εργασίας, ακριβώς υπό το φως αυτών των ε, νέων δημογραφικών μεταβολών τι μπορούμε να κάνουμε για να πετύχουμε τη συνέχιση προσφοράς εργασίας, θέσεων εργασίας για άτομα μιας κάποιας ηλικία και πώς ε, θα παροτρύνουμε για την εξέταση αυτών των ε, σημείων από στρατηγικής πλευράς. Να πείσουμε ότι είναι προς το συμφέρον όλων τα ηλικιωμένα άτομα να παραμείνουν απασχολούμενα και να έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο δράσης για τα ελικμένα άτομα και αυτό λοιπόν θα συζητηθεί από μας ε, με οποιαδήποτε προοπτική δημογραφικής αλλαγής ε, στην Ευρώπη. Σαφώς ε, η απασχόληση ατόμων πέρα από μια κάποια ηλικία, αυτή επαναλαμβάνω θα εξεταστεί όχι από μια και μόνο προεδρία αλλά και από τις επόμενες και κατά τη διάρκεια της περίοδου των έξι μηνών μας θα θέλαμε πάνω απ' όλα να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα της διάκρισης κατά των ατόμων αυτών, των ηλικιωμένων που είναι κοντά δηλαδή στην ηλικία συνταξιδότησης ή που την έχουν ξεπεράσει. για να δούμε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η Αντιπρόεδρος υπέβαλε ένα ερώτημα σχετικά. Έχουμε ένα σχέδιο οδηγίως που υποβλήθηκε τον Ιούνιο φέτος από την Επιτροπή και κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας ε, έχουμε σαν πρόθεση να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας πάνω σε αυτό το σχέδιο οδηγίας. Μπορώ να σας πω ότι στις 15 και 20 Ιουλίου η ομάδα εργασίας για κοινωνικά θέματα, η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό, θα συναντηθεί, θα συνεδριάσει και θα ασχοληθεί με αυτά τα σημεία και οι εργασίες δε αυτές θα συνεχιστούν το Σεπτέμβριο. Για τις οδηγίες αυτές επιθυμούμε να σημειώσουμε την ε, καλύτερη δυνατή πρόοδο μέχρι το τέλος της χρονιάς και ελπίζουμε ότι το θέμα αυτό θα αποτελέσει σημείο εξέταση στη μέση διάταξη του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ που θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου του 2011. Και αν τα πράγματα πάνε καλά, θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη μια έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά από τη γενική αυτή προσέγγιση, αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν αποτελέσματα της, των συναντήσεων της ομάδας αυτής της εργασίας που θα συνεδριάσει τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Να πάμε τώρα στον ελάχιστο μισθό, στην ελάχιστη αμοιβή, στο ελάχιστο εισόδημα. Είναι θέμα που είναι της αρμοδιότητας των κρατών μελών βέβαια αλλά μην ξεχνάμε την κινητικότητα των εργαζομένων και των εργοδοτών αλλά και των πολιτών που δεν εργάζονται ατόμων που επιλέγουν μετά τη συντεξιδότησή τους να ζήσουν σε άλλη χώρα από την μέχρι τότε, να δούμε πώς θα προστατευθούν κοινωνικά. Ποια είναι η άποψή μας ότι εκείνοι που έχουν εργαστεί και που έχουν ε, πληρώσει τους φόρους τους ε, σε οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να προστατεύονται κοινωνικά χωρίς διακρίσεις σε οποιοδήποτε κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Ε, τα τελευταία που είπατε θα τα γράψουμε σε μάρμαρο, θα τα σκαλίσουμε σε μάρμαρο στα χρονικά της Επιτροπής αυτής. Λοιπόν, Πλόμ και μετά σκητεύσα. Η κυρία Πλόμ πρώτα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι ενδιαφέρομαι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι σημαντικό μέσα ώστε τη μεταρρύθμιση των αγορών της απασχόλησης. Αυτή είναι η ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης κατά πόσο πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε επενδύσεις στην ε, εκπαίδευση για τις νέες αρμοδιότητες που χρειάζονται σήμερα, τις νέες ικανότητες των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκριτέψα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δύο σύντομε ερωτήσει, γιατί ξέρω δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Στο ανακοινωθέν τη ε, Επιτροπή για το Πολιετέ ε, ε, Δημοσιονομικό Πλαίσιο υπάρχουν διάφορε ενδιαφέρουσε πτυχέ και δεν θέλω να ξέρω ποια είναι η στάση τη Πολωνική Προεδρία. Δεύτερον, Θεωρείτε ότι είναι μια αποτελεσματική και χρήσιμη αυτή ε, μέθοδος ε, της ε, χρήσης των πόρων, δηλαδή το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ και Φραν είναι η, ε, η μας. Θα έχετε αργότερα την απόψη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω μια ερώτηση για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πώς θέλετε να εργαστείτε όσον αφορά τις ε, απαιτήσει ε, ε, σχετικά με την εκπαίδευση που αποκλείει τους νέους αυτή τη στιγμή και δεύτερον πώς θα μας βοηθήσετε για να φροντίσουμε ούτως ώστε ευρωπαϊκό επίπεδο τα χαμηλά επίπεδα ικανοτήτων να δουν να αυξάνεται το επίπεδο τον οικοδομητών αυτό για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις απασχόληση. Αυτή ήταν η ερώτηση τη κύρια Πλάμ. Ευχαριστώ. Κύριε Κουτιέρες, η δική σα ερώτηση προς ποιον απευθύνεται. Ωραία. Η κυρία Γεσλαβίσκα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω την ερώτησή μου στην Υπουργό κ. Μιανκόφσκα. Είπατε ότι η Πολωνική Προεδρία θα προτείνει ε, μία πιο συγκεκριμένη πτυχή, εδαφική πτυχή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δεκάδες χιλιάδων θέσεων απασχόλησης. Ποια είναι τα επικίνηματα για να υιοθετήσουμε αυτή τη διάσταση στο Ταμείο. Μήπως μπορώ να υποβάλω και μία ερώτηση του κ. Κοσλόφσκι που δυστυχώς χρειάστηκε να βγει από τον κύριο Κοσλόφσκι προς την κυρία Φέντακ. Όχι, όχι, όχι στην κυρία Φένταξ, στην κυρία Βιενκόφσκα προφανώς ήθελα να πω. Ερώτηση του κυρίου Γιάνν Κοσλόφσκι προς την κυρία Μινκόφσκα. Υπάρχουν πραγματικά πρόοδοι στις διαπραγματεύσεις το ώστε τα τέλη του 2011 τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να έχουν αρκετέ πληροφορίες για να αρχίσουν να διαπραγματεύουν τις ε, συνθήκες για τις εταιρικέ σχέσεις. Ευχαριστώ κύριε η Δική σας ερώτηση προς ποιον απευθύνεται. κύριε Υπουργέ, μπορείτε να πάρετε λόγο να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Όταν βλέπουμε στα διάφορα προγράμματα να αναφέρονται και άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες, ειδικά για το κοινωνικό ταμείο, τελικά βλέπουμε η κάλυψη να είναι πολύ περιορισμένη παρόλα όλα αυτά. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να κάνει καλύτερη στοχοθεσία ούτως ή άλλως. Όπως ε, έλεγα προηγουμένως, πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τις δραστηριότητε του Ταμείου αυτού και ως Προεδρία θα εντοπίσουμε μια σειρά στόχων προκειμένου να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες των... Ε, μάλλον να δούμε και τις... Ε, τα όσα χρειάζονται για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η Πολωνική Προεδρία θα ασχοληθεί μάλιστα με την ανάληψη πρωτοβουλειών στα πλαίσια αυτού του προπολογισμού. τρέχοντα την Πολωνική Προεδρία και με του υπεύθυνου τη Πολωνική Προεδρία, κάνουμε μια σχετική συζήτηση, ώστε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εκταμιεύσουμε κάποια κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπέρ των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε. Για την ερώτηση τη κυρία ε, Τιτλεύσκα και τη κυρία Πλάμπ, να είμαι σύντομη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και την επισητιστική βοήθεια. Το θέμα αυτό είναι τελείως καινούριο, όπως είπα. Πρέπει πρώτα να το μελετήσουμε, να επαληθεύσουμε κατά πόσον αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν υπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην ε, παγκοσμιοποίηση ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό θα απασχολήσει κατά πρώτον την ε, Πολωνική Προεδρία και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, όπως έλεγα, επιθυμούμε απλούστευση της πρόσβασης σε αυτό το ταμείο, κατά πρώτον. Έπειτα, μας ενδιαφέρει να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ υποβολής αιτήσεων και πρόσβασης, ε, απεμπλοκής τέλος πάντων των κονδυλίων. Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στις εκκλήσεις που μας απευθύνονται ως προς αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό θα δείξουμε κατά την απαραίτητη προσοχή. Το ερώτημα για την αδερφική διάσταση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις με την πολιτική συνοχή. Μόνον με προσαρμογή Τη απόδοση δημοσίων κονδυλίων στι τοπικέ ανάγκε, μπορούμε να ελπίζουμε ότι μια συγκεκριμένη περιοχή θα εκμεταλλευτεί το δυναμικό τη. αυτό που διαθέτει και θα ξεπεράσει και τα όρια τη Με την καλή έννοια. Αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί ξέρουμε ότι μιλούμε πολύ συχνά για δείκτες, για μέτρηση της πρόοδου. Η πρόοδος λοιπόν είναι ένα θέμα ευαίσθητο. Και επαναλαμβάνω, η διάσκεψη που θα οργανωθεί το Σεπτέμβριο σχετικά είναι πολύ σημαντική για μας. Και για να παραμείνω στην εδαφικότητα. E, Θέλουμε εδώ πραγματικά να φτάσουμε σε αυτούς που έχουν την ανάγκη μας. Για να παραμείνω στο παράδειγμα της Πολωνίας που γνωρίζω καλύτερα, Θέλουμε να φτάσουμε στις επιχειρήσεις, στις εταιρείε που σε τοπικό επίπεδο έχουν ανάγκη. Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την εκπαίδευση τώρα, να πω τα εξή. Το κοινωνικό ταμείο έχει για την ώρα εξαιρετικές ε, εμπειρίες. Για μας προτεραιότητα θα είναι να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση. Όμως καρπούς θα μπορούμε να δρέψουμε μόνο όταν απευθυνόμαστε σε μικρές ομάδες, μικρές εταιρείες, μικρές επιχειρήσεις και σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν τα ανάλογα εθνικά προγράμματα να συνδυαστούν με τη δική μας την ε, προσπάθεια και έπειτα να αποτιμήσουμε και την ε, αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέτρων. Η αποτελεσματικότητα του κοινωνικού ταμείου είναι κάτι που συχνά άλλωστε επικρίνεται. Εμείς θεωρούμε το ταμείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικότερα, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέλος, για την ερώτηση του κ. Κοζόφσκη. Ίσως επαναλαμβάνω τώρα πράγματα που τα είπα ήδη στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, όμως, εάν οι γενικοί κανονισμοί για τη λειτουργία των ταμείων υποβληθούν ως το Σεπτέμβριο, τότε μέχρι το τέλος του Πουρανικού Εξαμήνου το Δεκέμβριο μπορεί να έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για τα λειτουργικά προγράμματα. Ήδη έχει προβλεφθεί ένα χρονοδιάγραμμα σε συνδυασμό με τις επόμενες προεδρίες, την Δανέζικη και την Κυπριακή, ώστε η συζήτηση ακριβώς για τα προγράμματα εφαρμογής να αποτελέσει θέμα προτεραιότητας. Εδώ μα ενδιαφέρει το πού θα κατευθυνθούν τα κονδύλια, τι όροι θα τεθούν και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα μιλήσουμε και για το ring fencing, όπω είπα, τα μέτρα περί χάραξη των στόχων. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Η κυρία Κούντ νομίζω έφυγε. Η κυρία Στάιμπλουκ. Και ο κύριο Ντερόζα μετά. κυρία Στάιμπλουκ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Φέντακ, θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση του συναδέλφου Στιβενιού και την απάντησή σα. Πριν από δύο εβδομάδε ήμουν μέλο με στην προσπία των σοσιαδημοκράτων στο εργοτάξιο τη Φλαμονβέλ και είδαμε εκεί του όρου ε, διαβίωσης και εργασίας των αυσταλμένων εργαζομένων που είναι καταστροφικοί για μας. Μας είπανε ότι για φόρους και κοινωνικές ε, ε, εισφορές αφαιρούνται διάφορα ποσά από τους μισθούς των εργαζομένων αυτών. Δεν ξέρουμε τι γίνονται τα χρήματα αυτά γιατί δεν ήταν ούτε καν ασφαλισμένοι οι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν ή συμφωνείτε μαζί μας ότι χρειάζεται γι' αυτό μια νομοθετική ε, πρωτοβουλία για την αναθεώρηση της οδηγίας αποστολής εργαζομένων. Γιατί είμαι σίγουρη ότι μέχρι το τέλος των θερινών διακοπών μπορώ να σας δώσω πολλά περισσότερα παραδείγματα και από τη Γερμανία. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και με τους εργαζομένους δεν νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Τερόσα και μετά ο κύριος Νταρντέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, κυρία Φεντάκ, να σας υποβάλω μια ερώτηση όσον αφορά τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Αναφερθήκατε στην ε, συνοχή που θέλει να προωθήσει η Πολωνική Προεδρία, αλλά η ε, κοινωνική ένταξη είναι πάρα πολύ σημαντική για τη συνοχή και οι υπηρεσίες αυτές συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο συμφώνησε να υπάρχει το Γενάρη ένα νέο φόρουμ για τις κοινωνικές αυτές ε, υπηρεσίες. Σκοπεύει η Πολωνική Προεδρία να βοηθήσει στην προετοιμασία αυτού του φόρουμ. Ευχαριστώ. Ταρντέν και μετά Βουτιέρος Πρέστο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, να πάω στο θέμα της ε, μάχης ακριβώς, τη βάση αυτή, της μάχης κατά της φτώχειας. χαίρομαι γιατί τη σημασία σε αυτή τη βάση και θέλετε να υπάρξει αυτή η συζήτηση και μετά τη Κρακοβία κλπ. Και, και χαίρομαι και για κάτι άλλο. Και αυτό έχει να κάνει με τις δύο υπουργούς, ότι η επιστημική βοήθεια στους φτωχότερους θα βρει τρόπο επίλυσης της επόμενους αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην είναι εις βάρος άλλων κοινωνικών πολιτικών και για τη βάση αυτή και πάλι συζητάμε αυτή την έκθεση και θα πρέπει την ίδια στιγμή με τη σύμβαση στην Κρακοβία να ψηφιστεί. Υπάρχουν λεπτά θέματα τα οποία εξετάζονται. Το ελάχιστο εισόδημα και από ό,τι είδα ήταν μάλλον θετική αντιμετώπιση. Γι' αυτό πέστε μου ποια είναι η θέση σας και σε άλλο λεπτό θέμα πώς η οδηγία κατά της οριζόντιας διάκρισης θα μπορούσε να ισχύσει που κάτι που παγώνει σε επίπεδο συμβουλίου προς το παρόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και ο Γκουτιέρες ε, και κυρία Μωρέν πιο σύντομα ακόμα. Κύριε Γκουτιέρες, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ στην ε, κυρία Υπουργό για την παρουσία της στην Επιτροπή μας και τα όσα μας είπε. Ακριβώ έχουμε πρώτες ε, αναπτύξεις ιδεών. Μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, για την ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη, για να βγούμε ακόμα ισχυρότερα από την κρίση που η ελεγγύη αυτή θα πρέπει να έχει να κάνει με την πολιτική και με διάφορες χειρονομίες όμως και μου προκάλεσε κάποια έκπληξη, κάτι που είπατε στην αρχή της παρέμβασής σας ότι δεν σας αρέσουν αυτές οι αντιδράσεις στον κοινωνικό διάλογο αλλά ίσως και δεν μου αρέσουν εμένα τα κίνητρα που από τα οποία ξεκίνησαν αυτές οι εκδηλώσεις, αυτοί οι ε, διαδηλωτές, που είναι εργαζόμενοι και δεν καταλαβαίνουν τους λόγους της κρίσης. Ε, δεν καταλαβαίνουν επίσης ότι μερικές φορές αυτές οι λύσεις αντιμετώπισης της κρίσης ε, είναι ακριβώς οι απαιτήσει των ίδιων που προκάλεσαν την κρίση. Κάτι το συγκεκριμένο. Ναι, σίγουρα Χρειαζόμαστε καλύτερη πολιτική, πιο φιλόδοξη σχετικά με το ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο και την απασχόληση και έχουμε και επίσης προβλήματα για τους νέους, για εκείνους πάνω των 45 ετών, εκείνους με φυσικά προβλήματα, πώς ακριβώς ε, η πολιτική η Πολωνική Προεδρία θα αντιμετωπίσει το θέμα. Τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει στο Συμβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή για τα άτομα αυτά. Ευχαριστούμε κυρία présidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά την ερώτηση που έθεσε η Αντιπρόεδρος μας η κυρία Λίν. Είπατε για τα μαγνητικά πεδία και τη σχετική έκθεση ότι θέλετε να υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Σήμερα απέχουμε από αυτό το στόχο, Όμω ξέρουμε ότι υπάρχει και καταληκτική προθεσμία τον Απρίλιο. Ήθελα λοιπόν τη δική σα τη θέση για την χρήση των ε, κυμάτων αυτών για ιατρικούς σκοπούς. Στον τομέα της υγείας τα χρειαζόμαστε τα κύματα. Ε, ποια η θέση λοιπόν της Πολωνικής Προεδρίας. Ξέρουμε ότι στην εγκύκλιο του 2004 και τους σχετικούς κανόνες αποκλείονταν τα μέσα αυτά. Και δεδομένης σήμερα στις χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε και του χρονοδιαγράμματος που υπάρχει, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να ελπίζουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Τι λέτε. Κυρία Υπουργέ. Odpowiadając jeszcze raz na kwestię tego, co wydarzyło się we Ναι. Αυτό που ρωτήσατε σε σχέση με την Γαλλία και η αναθεώρηση της οδηγίας αυτής απαιτεί μια συμφωνία και με, τα, με τους κοινωνικούς εταίρους. Και με εκείνους θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα Πρέπει να εγγυηθούμε και καλέ συνθήκε εργασία ακόμα και σε παρόμοιες συνθήκε. Σε, παρόμοιες, σε τέτοιες περιστάσεις μάλλον. Ε, εδώ το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα κενά της οδηγία. αλλά και παράνομε δραστηριότητε πολλές φορές που υπάρχουν. Αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο επίσημη έρευνας και καταδικών. Εάν κάποιος καταχραστεί χρήματα, ή πάρει κονδύλια τα οποία μετά δεν τα χρησιμοποιήσει για νόμιμους σκοπούς, λογικά διώκεται και καταδικάζεται. Άρα, εν μέρη τουλάχιστον, το να αναλυφθεί δράση από τα αρμόδια όργανα είναι μια λύση. Και να είναι και ένα παράδειγμα για άλλα όργανα. Για τη συμμετοχή τώρα των κοινωνικών εταίρων να πω ότι ίσως την διαδικασία των νομοθετικών ε, μεταρρυθμίσεων να συμμετάσχουν περαιτέρω η κοινωνικοί ακριβώ εταίρεια για να βελτιώσουμε τα επίπεδα προστασία των ε, εργαζομένων και των δικαιωμάτων του. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του διαλόγου με του κοινωνικού εταίρου. Και βεβαίω και μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερε προτάσει του. Έγινε λόγος και για διάφορε διαδηλώσει κατά τη διάρκεια των ε, ερωτήσεων. Μα προφανώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρήζουν ε, εθνικής μέρημνα περισσότερο από ότι ευρωπαϊκή. Αλλά ο κοινωνικός διάλογος ε, πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Διότι Υπάρχει κόσμος που κατεβαίνει στο δρόμο ε, για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν δείχνουν καλή διάθεση για να οργανωθεί διάλογο, συζήτηση επικοδομητική μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων λόγου χάρη, τότε ο κόσμος θα διαμαρτυρηθεί, θα αγανακτήσει. Γι' αυτό λοιπόν παρατρένουμε του κοινωνικού εταίρου να εκφράζονται. Να εκφράζονται ω το δυνατόν πιο ανοιχτά και με μεγαλύτερη σαφήνεια. Προκειμένου να βρεθεί συμφωνία η οποία θα μπορούσε να αποτελεί βάση κοινωνικής σύμβασης. Αυτό για να συμβεί πρέπει να υπάρχει προφανώς και πρόσφορο έδαφος. Διότι τι συνέπειε τη κρίση όλοι θα τι απομισθούν. Και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και βεβαίω όσοι έχουν πληγεί περισσότερο. Αλλά εδώ μιλάμε για στοιχειώδη δικαιοσύνη πλέον. Μερικές αποφάσεις είναι σκληρές, αλλά μπορεί να είναι δίκαιες και ισότιμες για όλους τα αποτελέσματά τους. Γι' αυτό λοιπόν κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, κάθε ένωση εργαζομένων έχει δικαίωμα να απεργήσει, έχει δικαίωμα να εκφράσει τι απόψει του. Αλλά πολύ καλύτερα θα ήταν να υπήρχε μια συμφωνία. Και μάλιστα εκ των προτέρων ώστε να αποφευχθεί αυτού του είδους η ένταση την οποία ζούμε σήμερα. Πρέπει να δοκιμάσουμε, να συμφωνήσουμε εξ αρχής, ώστε να μοιράσουμε εξίσου τις συνέπειες και τις δυσκολίες που προκαλεί η κρίση. Τώρα, κάτι ακόμη που θα το συζητήσουμε τουλάχιστον άλλες δύο φορές, πρώτα απ' όλα στην πλατφόρμα κατά τις φτώχειας, διάσκεψη πολύ σημαντική τον Οκτώβριο στην Κρακοβία, όπου θέλουμε να επισκοπήσουμε εκεί. το πώς έχουν ελοποιηθεί δράσεις που αποφασίστηκαν στα πλαίσια των, της πλατφόρμας για τον περιορισμό του κοινωνικού πολιτισμού και την καταπολέμηση της στόχης. Προσκαλούμε όλους τους βουλευτές και τις βουλευτές φυσικά που ενδιαφέρονται να έρθουν στην Κρακοβία για να συμμετάσχουν σε αυτή τη ε, διάσκεψη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα παιδεία. Όχι, προηγουμένως, ναι, ναι, ε, το θέμα του κατά πόσον θα συμπεριλαμβάνονται τα κύματα ή όχι. Νομίζω η οδηγία πρέπει να εγγυάται την προστασία όλων των εργαζομένων. Πρέπει οι διαπραγματεύσει μα να πάρουν τέτοια κατεύθυνση ώστε όλοι οι εργαζόμενοι που είναι εκτεθειμένοι στο ελάχιστο στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία προστατεύονται παρκώ. Ίσως να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα πριν το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Με λίγη καλή θέληση ίσως τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. E, λοιπόν, το θέμα ερωτήσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, κοινού ενδιαφέροντες. Τι παρατηρούμε ότι όλοι οι συμμετείχοντες, ε, όλοι που παρέχουν αυτές τις ε, υπηρεσίες, όσοι τις χρησιμοποιούν, τα κράτη-μέλη, όλοι ενδιαφέρονται για καλή ποιότητα αυτών των υπηρεσιών και υπάρχει ένα πλαίσιο, μια κατευθυντήρια γραμμή η οποία μας δείχνει πώς θα υπάρξει αυτή η καλή ποιότητα, πώς θα ισχύσουν οι προδιαγραφές οι με πρωτοβουλία που προέρχεται από μία στρατηγική η οποία καλύπτει και τη χρηματοδότηση στη βάση των κοινωνικών προγραμμάτων και το Σύμβουλο ΕΠΣΚΟ υιοθέτησε το σχετικό κείμενο το 2010 και οι κατευθυντήριες γραμμές ε, υιοθετήθηκαν σαν συμπεράσματα του Συμβουλίου και επίσης ένα φόρουμ για τις υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντες και εμείς συμμετέχουμε στην προετοιμασία αυτής της συνάντησης που θα διεξαχθεί την επόμενη χρονιά και σας προσκαλούμε και στις προετοιμασίες και στι εργασίε. να συμμετάσχετε. Ναι. θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Εξ ονόματο λοιπόν όλων των συναδέλφων, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και να σας βεβαιώσω ότι τα μέλη της Επιτροπής μας είναι στο πλευρό σας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θέλουμε η Προεδρία σας να γίνει ακριβώς η κατάλληλη ευκαιρία ώστε για να επιτύχουμε του στόχου των οποίων έχει τα την ευθύνη. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. pendant que les ministres nous quittent, je voudrais euh, donner euh, la parole. Τώρα που φεύγουν οι υπουργοί, δεν θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιολίχ για την παρουσία του ΣΥ των τροπολογιών για την έκθεση, για την ε, και Η ανατομία της ευρωπαϊκής αγοράς, τον συλλογισμό μάλλον της ευρωπαϊκής αγοράς, της πολιτικής δημοσίων συμβάσεων και ψηλεύσεων. Η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο. Madame Girling. Euh, Με συγχωρείτε, έκανα λάθο. Γιατί πριν το σημείο τη κυρία Γκέρλινγκ πρέπει να εξετάσουμε και το σημείο 5 την ε, καταπολέμηση του θετουμένου τη πρώτης εγκατάλειψης του σχολείου. Ζητώ συγγνώμη την κυρία Κιόλη και θα ήθελα να σα δώσω το λόγο για την παρουσίαση των τροπολογιών κυρία Χίρς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, του σκιώδες συγητές και συγγήτρες για την καλή συνεργασία πάνω σε αυτό το θέμα. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε μια συνεδρίαση εξετάσαμε τις πολλές τροπολογίες που υποβλήθησαν. 125 τροπολογίες υπήρχαν, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές, πολύ ενδιαφέρουσες και έτσι διευκρινίζουν πολύ καλύτερα τον τομέα. Αλλά νομίζω ότι μια που είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα, όπως η πρόεδρε του σχολείου, χρειάζεται πραγματικά να περάσουμε στις λεπτομέρειες. Προσπαθήσαμε αυτές τις 25 τροπολογίες να τις ενώσουμε κάπως. Για 50 τροπολογίες το καταφέραμε. Καταλήξαμε στις συμβαστικές τροπολογίες που τις έχετε μπροστά σας. και για τις οποίες μέχρι στιγμής ε, άκουσα μόνο στην ενετική ε, τοποθέτηση από όλες τις πολιτικές ομάδες, για τις συμβαστικές τροπολογίες δηλαδή και από εκείνου που υπέβαλαν τις τροπολογίες. Καλά προχωρήσαμε νομίζω. Βέβαια υπήρχαν και επικαλυπτόμενες τροπολογίες που μπορούσαμε να συνενώσουμε. Βέβαια το κάθε σημείο τώρα είναι πιο μακρύ από ό,τι τα προηγουμένα, αλλά όπως σας είπα το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δικαιολογεί νομίζω να, ένα ξε... να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα κράτη-μέλη. Πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για μας. Χαίρομαι που βρήκαν τόσο πολλές ε, τροπολογίες. Παρουσίαση των ε, κρατών μελών και των εθνικών προγραμμάτων ε, πανέρχεται εδώ σε εμά στην αρμόδια επιτροπή. Δυστυχώ βέβαια όσον αφορά το θέμα αυτό, αρμοδιότητα δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα κράτη-μέλη. Εξαρτάμεθα λοιπόν από τη συνεργασία μαζί του. Και χαίρομαι που τα κράτη-μέλη μέσω τη Κομισιόν μπορούν σε ένα χρόνο να μα παρουσιάσουν τις επιτυχίες τους. Πολύ καλό αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και για τις προσθήκε να τονίσουμε ότι πρόκειται για θέμα χρηματοδότηση σαφές αυτό. Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης βέβαια σε ορισμένες χώρες έχουν περιοριστεί λίγο ή και περισσότερο οι προπολογισμοί για την παιδεία και αυτό είναι μια σημαντική πτυχή που έχει συμπεριληφθεί στη συμβαστική τροπολογία Α. Και αυτό πάλι είναι ένα μήνυμα. Λέμε στα κράτη-μέλη προσέξτε το αυτό το σημείο αυτό. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα βέβαια. Ένα άλλο θέμα αφορά τους Ρωμά, τα παιδιά των Ρωμά. Αυτό ήταν καταρχήν ένα σημείο συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι σε συσχετισμό με το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε το θέμα αυτό πολύ εις βάθος και ότι αποφάσαμε και μία στρατηγική για τους Ρωμά. Είναι σωστό τώρα αυτό να το κατοπτρίσουν στις διάφορες μας χρονοποδοτήσεις. Να μην πούμε είχαμε αποφασίσει κάποια πολιτική του Ρωμά που αποφασίστηκε τότε και είναι καλό να αντικατοπτρίσετε τώρα παντού και αυτό μου φαίνεται ότι είναι καλό που βρήκαμε μια πολύ ωραία συμβαστική τροπολογία γι' αυτό. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που λήφθαν υπόφθη, το θέμα της εκπαίδευσης των διδασκάλων, Πώς θα γίνει αυτό το αναφέρουμε μόνο η παρόδο η Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων εξετάζει τις λεπτομέρειες. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τις διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας και να υπάρξει ιδιαίτερα μάθημα για κάποιους μαθητές. Αυτό υπάρχει στην ε, ε, Τροπολογία τάφ, συμβαστική τροπολογία τάφ. Επίσης αναφερόμαστε ότι αυτό αφορά πιο πολύ τους, ε, τα γόρια από τα κορίτσια. Και νομίζω ότι έχουμε ε, μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης όταν τελικά ψηφίσουμε πάνω στην έκθεση. Αυτά από μέρους μου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τους συσκευοσυγητές για την καλή συνεργασία και με χαρά θα ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Πρώτα, εγώ σας ευχαριστώ. Θα παρακαλώ τους ομιλητές να είναι πολύ σύντομοι. Γιατί έχουμε δυστυχώ πάρα πολύ βεβερμένη μέσα διάταξη. Μου φαίνεται ότι όλο το ίδια λέω. Ανακοσα και μετά κύριος Κουτσιέρες Πρίτο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Εγώ επέφερα μία τροπολογία που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αλλά δεν είναι αυτό, αυτό που θέλω να αναπτύξω, γιατί διαβάζοντας τροπολογίες μπορώ να συμφωνήσω με τις περισσότερες από αυτέ. Και θα ήθελα να τονίσω ε, ιδιαίτερα κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν πάνω στις κατηγορίες. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες σε κάθε κράτος μέλος και έτσι δεν μπορέσουμε να προχωρήσουμε εκτός εάν έχουμε μία ομοιόμορφη αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Γκουτιέρη Πριώτο. Κύριε Πρόεδρε, γρήγορα, γρήγορα. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί έδειξε κατανόηση σε μια έκθεση γνωμοδότησης αλλά σημαντικό για μένα για την Επιτροπή μας, γιατί οπωσδήποτε η εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες και όσο καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση έχει κανείς, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει και λιγότερος κοινωνικός ε, επαγγελματικός αποκλεισμός. Είναι λοιπόν σημαντικότατο για μένα για το μέλλον το κοινωνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και νομίζω ότι η εργασία ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτή την ε, έκθεση με τις συμβασικέ τροπολογίες, τις οποίες πετύχαμε όλες οι ομάδες, με κάτι το περισσότερο ολοκληρωμένο, το περισσότερο φιλόδοξο, που έχει να κάνει και με την ε, πρόβλημα ακριβώ της εγκατάλειψης του σχολείου ε, και την κατάσταση την εργασιακή, την οικογενειακή, το πώς σε διάφορα κέντρα εκπαιδευτικά μπορεί κανείς να συμβιώσει, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς, πώς μπορεί να βελτιωθεί το όλο σύστημα, ξεκινώντας από την καρδιά του συστήματος που είναι οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και κρίμα που στα συμβαστικά αυτά δεν μπορούσαμε να συμπεριλάμε και μια σημαντική για μας τροπολογία η οποία όμως δεν πέρασε. Θα ήθελα να σας πω Ποια είναι η φιλοσοφία της, ε, μια αύξηση στην ε, δημόσια ακριβώς επένδυση για τη βελτίωση αυτού του συστήματος για ένα λόγο απλό ότι είναι και εκεί ο κεντρικός πυρήνας είναι αυτή η πολιτική ανακατανομής για ένα δημόσιο σύστημα που επέτρεψε τη δημιουργία μιας μέσης τάξης ευρωπαϊκής ισχυρής εδώ σε αυτή την περίοδο κρίσης η βελτίωση και της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης κυρίως της δημόσιας είναι ο καλύτερος τρόπος η βοήθεια βοήθεια προ αυτού για να ξεφύγουν από την κρίση. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τι προσπάθειε που κατέβαλε για την εργασία τη ακριβώ ε, στα πλαίσια αυτή τη ε, έκθεση νομοδότησης και για τι συμφωνίε τι οποίε πέτυχε με τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Και μετά το Μασμάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα... Θέλω να είμαι σύντομο γιατί το προτείνεται αυτό ένα θέμα που συζητήσαμε ήδη για μακρόν ε, το θέμα αυτό της πρόσφυγας κατά σχολείο από όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε γρήγορα όσον αφορά την ανάλυση του φαινομένου και οι πολλές ε, τροπολογίες που βρήκαν και οι συμβαστικές τροπολογίες που επιτεύχθησαν κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την καλή συνεργασία με τους πιο ηγητές δεν είχαμε κανένα πρόβλημα εκτός από τη συμβαστική ε, Β. Αυτή η συμβιστική τροπολογία αφορά τους Ρωμά και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, να ψήφισαν σε κάποιον τομέα αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε, ε, να χρησιμοποιούμε αυτές τις ε, διατάξεις για τους Ρωμά παντού, οριζόντια. Με αυτό το σημείο δεν μπορούμε απόλυτα να συμφωνήσουμε λοιπόν, αλλά γενικά η πρόκειται για μια πολύ καλή έκθεση που θα τύχει σίγουρα ευρεία συνένεση. Και τελειώντα, ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία και για την καλή έκθεση που πέτυχε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Κύριο Τόμα Μαν. Και μετά κύριο Τουρινέ. Μπερδεύομαι. Ο κύριο Σουμάν και η κυρία Τούρνεν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον, η οποία μας είπε ότι ήταν πολύ καλή συνεννόηση με τους πρώτους εισηγητές. Υποθέτω ότι έλαβες και τις τροπολογίες με τα ονόματα των προτινόντων, γιατί βλέπουμε στις συμβαστικές σου λύσεις ότι παρά τις κάποιες διαφωνίες βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο μήκος σχήματος. Πολύ καλά λοιπόν φαίνεται ότι θα αντιμετωπιστεί το, ζήτημα αυτό, ιδίως ό,τι φορά τις εξαιρέσεις. Δεν πρέπει να είναι θέμα μόνο των ε, γονιών ε, κατά πόσο θα έχουν ευκαιρίε τα παιδιά στη ζωή τους ή όχι. Αλλά ακριβώς πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτό το θέμα της, έγκυρης εγκατάλειψη, της πρόορης εγκατάληψης. Ε, είχαμε 125 τροπολογίες, πολύ καλό αυτό, οι συμβασμοί ήταν πολύ καλοί και χαίρομαι ότι το θέμα των Ρωμά, όπως είπε ο είναι ξεχωριστό θέμα. Δηλαδή θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη μας, να βγούμε από τις γενικές ε, διακηρύξεις και να έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και χαίρομαι που πετύχαμε αυτόν τον συμβιβασμό. Πολύ καλή έκθεση λοιπόν. Θα ήθελα όμως, πρόκειται πάλι για μια έκθεση τροπο, ε, ε πρωτοβουλίας και θέλω κάπου να εξεταστεί και να μην καταλήξει να συζητηθεί στο Στρασβούργο τη Δευτέρα στις 12 παρατέρα του νύχτα και να μην ακούσει κανένα να μην καταλάβει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε γιατί περιμένουν όλοι οι άνθρωποι να μας ακούσουν, οι πολίτες να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι συγκεκριμένο. Συγχαίρω λοιπόν τους πάντες και ιδίως την αγαπητή Νάντια. Øh, øh, Κυρία Πρόεδρε, Εξ ονόματος των Πρασίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άντια Χίρς για την άριστη αυτή συνεργασία. Ναι, πραγματικά μας ικανοποιούν αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες. Τόμας Μαν, τι είπε, ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να έχει μια καλή θέση στην Ολομέλεια και στη διάσκεψη των Προέδρων ίσως θα διαφωνεί. Πάντως πρόκειται για κάτι το συγκεκριμένο, για μια πραγματική βοήθεια στη στρατηγική του 2020. Και ένα σχόλιο στο πρώτο πρόγραμμα αυτό σε εθνικό επίπεδο κανονικά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε καλή περίοπτη θέση. Λοιπόν, Εάν επιθυμούμε στην Ευρώπη να δώσουμε τη μάχη μας κατά του αποκλεισμού, του σχολικού, της εγκατάλειψης, της εξόδα το σχολείο και είναι και ο καλύτερος τρόπος για τη μάχη μας κατά του αποκλεισμού, της φτώχειας. Είναι η ευκαιρία να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Είναι ο καλύτερος τρόπος να εγγυηθούμε την μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και επίσης κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι και η κοινωνική διάσταση της οικονομίας. Χαίρομαι. Είμαι ευτυχισμένη γιατί εδώ δείχνουμε σταθερή θέση απέναντι στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε πάντα να εφιστάμεθα τις μειώσεις του προπολογισμού των κονδυλίων στην εκπαίδευση. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια πραγματική καταστροφή. Δύο πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Υπάρχει ένα νέο πρόβλημα ανάμεσα σε νέους άνδρες και γυναίκες. Τα νέα παιδιά, τα νέα αγόρια είναι εκείνα που εγκαταλείπουν το σχολείο και αποτελούν μια υποκατηγορία κατά κάποιο τρόπο. Και είναι σημαντικό να το επισημαίνουμε αυτό. Μιλάμε πολύ συχνά για τα προβλήματα των γυναικών ε, και για ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Εδώ έχουμε ε, καταρνητικό από την άλλη πλευρά για τους άνδρες. Εντάξει δεν θα καταχραστώ του χρόνου μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για άριστη έκθεση. Πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Μετά από όλα αυτά τα εγκόμια έχετε πάλι το λόγο για να απαντήσετε αν θέλετε. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ για όλα αυτά τα θετικά που άκουσα. Θα χαιρόμουν λοιπόν πραγματικά, εάν δεν εξετάσουμε μετά τις 11 τη Δευτέρα τη νύχτα στο Στρασβούργο την έκθεση αυτή, θα δούμε τώρα πού θα τοποθετηθεί. Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, ιδίω όπως ελεγχθεί ήδη, σε σχέση και με τη στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ίσως ε, αν δεν το θέσουμε σε καλή θέση στην ημερήσια δίδαξη για κοινωνικούς λόγους, ίσως για οικονομικούς. Τώρα, όσον αφορά τους δείκτες που μέσα στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων δράσης ε, και της καταμέτρησης ε, της προώρης εγκατάλειψης, υπάρχει η τροπολογία 23 των σοσιαλιστών που ζητάνε ακριβώς την εισαγωγή των δικτών. Εάν υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την τροπολογία, ο στόχος είναι να συμφωνήσουμε πάνω σε κάποιους κοινούς δείκτες. θα ψηφίσουμε εμείς, η Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων θα εξετάσει το Σεπτέμβριο τη δική έκθεση. Έτσι έχουμε δηλαδή το χρόνο κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών να συζητήσουμε με του συναδέλφου στην Πολιτιστική Επιτροπή και το Σεπτέμβριο να ξανατοποθετηθούμε για την έκθεση αυτή μέσα στι επιτροπέ αυτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλοι οι που Ελπίζω να άκουσαν αυτό που ελέγχθη. Να υπάρχει δηλαδή καλή αντιμετώπιση όταν τεθεί στην μεσία διάταξη το θέμα. Περνάμε στο σημείο 6 μεσίας διάταξη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λούτβιξον για την εξέταση των τροπολογιών για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του Νομισμού των Οικονομικών Πολιτικών. Έχει το λόγο. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω του συναδέλφου, ιδίω του και εισηγητέ, διότι εδώ είχαμε μια πολύ πρόσφορη συνεργασία και κάναμε όλοι μεγάλε παραχωρήσει για να καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει. Μπορείτε σήμερα ήδη να δείτε τον κατάλογο με τι δικέ μου τι προτάσει. Από αυτέ θα συμπεράνετε ότι έχω προτείνει και κάποιε προφορικέ τροπολογίε ώστε να γίνουν κάποιες ε, ίσονο σημασίας διορθώσεις υπήρξαν τροπολογίες που ξεπερνούσαν την αρμοδιότητα ή μάλλον το πεδίο που αφορούσε η έκθεση αυτή, αλλά βρήκαμε λύσεις και δεν νομίζω ότι είναι πολλά τα προβλήματα που παραμένουν εκκρεμή. Απλώς μία πρόταση θέλω να αναφέρω και σε αυτή να σταθώ, η τροπολογία 63. Εκεί με κάθε σεβασμό, επειδή δεν συμφωνούμε φυσικά πάντοτε όλοι. Νομίζω ότι εδώ ξεπερνάμε κάπως το πεδίο της ε, ε, επιτροπής μας και της έκθεσης για το πώς διοργανώνεται η εργασία και η κοινωνική προστασία κυρίως των ανέργων. Εδώ νομίζω ότι υπονομεύουμε λίγο την αξιοπιστία της έκθεσης. Ακόμη και αν συμφωνούμε σε όλα τα υπόλοιπα. Το φάσμα που καλύπτει η έκθεση αυτή δεν αφορά το να διθετήσουμε το πώς τα κάτι μέλη έχουν οργανώσει την κοινωνική τους ασφάλεια και πρόνοια. Ως εισηγητής θα έλεγα να καταψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Βεβαίω έχετε την ε, ελευθερία να αποφασίσετε και να ψηφίσετε όπως νομίζετε. Όμως, ε, για τις δικές μου συστάσεις ε, όσον αφορά την ψηφοφορία, έχετε δει τι απόψεις έχω. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Είμαι ανοιχτό και στις δικές σας προτάσεις και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι έως την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι συμβαστικές λύσεις. Συμφωνώ με όλες. Νομίζω αυτό που φάνηκε από τις συμβαστικές λύσεις, το νήμα που διατρέχει όλε, είναι ότι θελήσαμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την Απασχόληση, με την έρευνα και την ανάπτυξη, με την ε, ε, ανάπτυξη και την ε, κατάρτιση, την επαγγελματική εκπαίδευση, τα προσόντα, τις δεξιότητες, επιδιώκουμε όλοι κοινού στόχου και βλέπουμε ότι και το Κοινοβούλιο έχει εδώ να δραματίσει έναν ενεργό ρόλο. Και πάλι να πω ότι στι συμβαστικέ λύσει έχουμε συμπεριλάβει και του ε, βασικότερου στόχου από την στρατηγική για την Ευρώπη το 2020. Πολύ σωστά έχουν ενσωματωθεί λοιπόν στο κείμενο. Νομίζω με τι προφορικέ τροπολογίε βελτιώνεται το κείμενο και θα συμφωνήσω μαζί σα ακόμη και στο θέμα τη τροπολογία 63. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βουλό. Και μετά ο κύριος Κομφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ξεκινάει ένα κύκλο σε συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και για να δημιουργηθούν σχέσει συνεργασία μεταξύ οικονομικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών πολιτικών στα κράτη-μέλη για την ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη, όπω προβλέπεται στη στρατηγική για το 2020. Εδώ λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Λίβιξον για την εξαιρετική του εργασία ω εισηγητή και του συναδέλφου που συνεισέφεραν σε αυτό το σχέδιο έκθεση. Να χαιρετήσω ιδιαίτερω ε, την προσπάθεια για τι συμβαστικέ τροπολογίε που πραγματικά το πνεύμα όλων των τροπολογιών που υποβλήθησαν με τρόπο πολύ σωστό ε, εκπροσωπείται, πράγμα που είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Δεν θέλω να περιοριστώ εδώ στο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου ω προ την στρατηγική ε, ή το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Απλώ να μπω σε λεπτομέρειε για κάποιε πολιτικέ που θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πέραν λοιπόν των τροπολογιών που προτάθηκαν, υπάρχουν δύο σημεία, τροπολογίε 63, στην οποία θα επανέλθω, και 69. Για την 69 αποφασίσαμε να αποσυρθεί. Είναι ένα σημείο που μας φάνηκε σημαντικό να θίγει, διότι δεν υπάρχει λόγο. ο αντίκτυπο τη οικονομική κρίση συγκεκριμένα και οι δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών να βαραίνουν μόνο τον Ευρωπαίο πολίτη. Λογικό βρήκα να υπάρξει και ο λεγόμενος φόρος των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και εκεί να ανατεθεί ένα μέρος της ευθύνης, του βάρους της κρίσης. Όχι όλα να τα απομίζονται οι απλοί πολίτες. Συνειδητοποιώ βεβαίω ότι ο φόρος αυτός των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι μια δημοσιονομική ε, ρύθμιση που δεν έχει αναγκαστικά τη θέση του εδώ. Γι' αυτό λοιπόν δεχτήκαμε ως ομάδα να αποσύρουμε την τροπολογία 69. Παραμένει όμως 63. Για την τροπολογία 63, για την οποία δεν καταλήξαμε σε συμβαστική λύση, να πω ότι στόχο έχει να προτείνει όλες οι υποκατάστατες καλύψεις τα επιδόματα για όσους ε, δεν είναι σε θέση να βρουν εργασία, σε περιόδους ε, κακής σοδιάς, ισχνών αγελάδων, θα πρέπει να ε, σκεφτούμε ότι βαρύνουν ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη. Ιδίω όταν δεν συνοδεύονται από μια σκόπιμη πολιτική απασχόληση. Δεν διανύουμε δυστυχώ μια περίοδο που μπορούν τα κράτη-μέλη να προβλέπουν και υποκατάστατα επιδόματα στους ανέργους, χωρίς να υπάρχει και κάποια ελπίδα για να αλλάξει κατάσταση άμεσα, για προοπτική απασχόληση. Την τροπολογία λοιπόν 63 ε, παρατρύνω να την υπερψηφίσουμε, ιδίω τα μέλη της ομάδας μου. Και επίσης για τις υπόλοιπες συμβαστικές λύσεις, όπως τις εγκρίναμε με τον κύριο Λίβινσον, πραγματικά συστήνω ε, θερμά του συναδέλφου να την εγκρίνουν. Ε, ο κ. Κοφεράτη. Και θα προσθέσω και εγώ κάτι, λέει ο Πρόεδρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, ε, άριστη εργασία του συγητού μαζί με τους κοιόδης συγητές. Αυτό που ιδιαίτερα θα ήθελα είναι να τονίσω αυτή τη ε, δυνατότητα, όπως το είπαμε, σε μια τροπολογία με τον συνάδελφο για την ενίσχυση του διαλόγου του κοινωνικού. Πώς ε, θα μπορούσε να έχει θεσμικό χαρακτήρα αυτή η επαφή μεταξύ της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων ε, και οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν ε, μέσω συγκεκριμένων καλά στοχευμένων εγγραφών να μπορέσουν να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν τις προτάσεις Επιτροπής να σταθεροποιήσουμε και να παγιώσουμε στο χρόνο αργότερα. Να το κάνουμε αυτό για να δώσουμε περαιτέρω όθηση στον κοινωνικό διάλογο. Διαφορετικά ποιος είναι ο κίνδυνος ε, να ε, γίνει κάτι το περιθερικό, κάτι το φτωχό. Να υπενθυμίσω επίσης κάτι για μια διαφή... διατύπωση παρόμοια που είναι στην ε, έκθεση για την κρίση που προχθές εγκρίναμε πολλά ε, λέγοντας αυτό και το συμμερίζονται και αρκετοί. Το καλό είναι πολλά μέρη να είναι μέρε των ε, συγκεκριμένων μεμονωμένων μέτρων των νομοθετικών ή των γνωμοτήσεων που θα υποβληθούν πάνω σε θέματα που μια αρμόδια επιτροπή συμπερίλαβε στι εργασίε τη ε, και να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένο χαρακτήρα σε ενδείξει εδώ στην έκθεση για την κρίση θα μπορούσαν να αποτελούν μόνο πολιτικέ ενδείξει. Εδώ όμω μπορεί να αποτελέσει κάτι, ένα συγκεκριμένο απτό στοιχείο και επιχειρησιακό μάλιστα. Σα ευχαριστώ. Ναι, μετά από όσο είπε ο Κοφεράτη, συμφωνώ και εγώ και να επανέλθω στο θέμα της 63 τροπολογίας, γιατί είναι η πρώτη τα μέλη εδώ της Επιτροπής που ανησυχούν ε, γιατί στον κοινωνικό τομέα αυτό το εξάμεινο το ευρωπαϊκό να έχουν όλη την εντύπωση ότι επί Επιτροπή στους κοινωνικούς εταίρους τους λέει ακριβώς και στην εθνική τους ακόμα νομοθεσία τι θα πρέπει να κάνουν. Τους υπαγορεύουν λοιπόν εδώ, ε, να ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία 63 του κ. Μπολάνου. Ε, εντάξει, όχι επί τη ουσία. Ορισμένοι θέλουν έτσι να ξεκινήσουν την όλη συζήτηση. Εμεί εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι γίνεται από τη μεριά, τι λέμε ότι όχι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να είμαστε στη μέση σε αυτά εδώ, στα επεξεργασία όλων αυτών, ούτε να λέμε στου γενικού εταιρείε τι πρέπει να κάνουμε και μετά να ψηφίσουμε ανθρωπολογία. Τι γίνεται, νομίζω ότι είναι απόλυτη αντίφαση αυτό και όλοι μας θα πρέπει να το σκεφτούμε εάν χρειάζεται μια παρόμοια τροπολογία. Ακόμα και ο ίδιος ο συντάκτης της τροπολογίας αυτής, ο οποίος νομίζω ότι κανονικά θα, μάλλον θα θέλει να αποσύρει τροπολογία για να γίνει αντικείμενο πολιτικής συζήτησης και την παράθεση στη χώρα του, αλλά όχι εδώ. Τέλο πάντων, για τι συμβαστικέ τροπολογίε έριξα με προσοχή μια κάποια ματιά εκεί να σας πω δύο πραγματάκια. Εντάξει, ανακατεύομαι με αυτό που δεν με αφορά, αλλά τι να κάνω, το είδα. Την ε, δέλτα τροπολογία. Για να μπορέσουμε να συμπεριλάμε πολλά πράγματα, ακριβώς αναφέρουν πολλά και διάφορα, αλλά υπάρχει μια μικροεπανάληψη που είναι εις βάρος ίσως μας ακριβώς για τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου και έχουμε, είναι η δεύτερη φορά που αναπτύσσεται, αναφέρεται το θέμα αυτό and the principle of this uh, και social dialogue uh, αυτό στο δεύτερο μέρος νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε at all level σε κάθε επίπεδο και the democratic accountability που χρειάζεται να εξασφαλιστεί σε κάθε επίπεδο. Αυτή είναι η τελευταία μου λοιπόν υπόδειξη και στο H το λατινικό. Ναι, καταλαβαίνω ότι θέλησατε να του να συμπεριλάβετε αυτήν την τροπολογία στο business sector του και αντιγόνης Παπαδοπούλου εδώ, αλλά νομίζω ότι αυτός ο business sector νομίζω ότι εκπροσωπούται Ήταν ε, να βάλουμε το να συμπεριλαμβάνει και τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εντάξει, καλά και οι δύο διατυπώσεις, αλλά μην μπούμε δύο φορές και οι εργοδότες και το business sector. Τι είναι, αυτή είναι η business sector. Οι εργοδότες. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Στο συνάδελφο Μπουλάν να του πω κάτι. Συμφωνώ ιδιαίτερα με την τροπολογία του την 69 και θα χαιρόμαστε πραγματικά να την υπερψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Αλλά καταλαβαίνω για ποιο λόγο απέσυρε την τροπολογία αυτή. Όλα αυτά τα επιχειρήματα για την 69 τα ίδια ισχύουν και για την τροπολογία 63 μιλάμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο αυτή τη διαδικασία και όχι για τις πολιτικές απασχόλησεις που άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Καθαρά θεωρούμε ότι αυτά δεν συμβιβάζονται με την όλη έκθεση. Τι γίνεται, μήπως είμαστε εκτός αρμοδιοτήτων μας. Είναι μια τροπολογία που δεν μπορεί να ψηφιστεί, γιατί εδώ δεν μιλάμε για την απασχόληση, μιλάμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, για τον κύριο δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να καταψηφίσω αύριο, αλλά πρόκειται για θέμα διαδικαστικό ίσως. Δεν θα πρέπει να ανακατεύουμε, να μπερδεύουμε το πάντα, γιατί δεν θα έχουμε ένα τελικό στόχο και σκοπό. Έτσι. Αυτό θα ήθελα να πω. Πρόκειται για ένα ε, θέμα κανονισμού εδώ, το να συμπεριληφθεί όχι αυτή η τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Ναι, Λούντβιξαν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μπολάν κάτι θα ήθελα να πει. Μισό λεπτό. Καλύτερα να τον ακούσουμε πριν από εσά. Για την τροπολογία 69. Είπα γιατί να αποσυρθεί. Αυτό ο φόρο και όλου ο μηχανισμό δεν, δεν είναι καλό σχεδιασμένο. σω δεν θα πρέπει τώρα να το θίξουμε ιδιαίτερα. Αλλά τώρα για το πώ αυτό ανακατεύεται με την κοινωνική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συστάσεις περί προπολογισμού στα κράτη-μέλη, εκείνα με τις περισσότερα ελλείμματα που αντιμετωπίζουν την κρίση, Μήπω μπορείτε να με εξηγήσετε πού είναι τα όρια της επικορικότητας εδώ, Νομίζω ότι παντού μπαίνουν αυτά σε κάθε πτυχή της ε, πολιτικής προϋπολογισμού στα κρατημένη. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει συστάσεις ε, για την ε, για τους φόρους, για τους μισθούς, για πολλά και διάφορα μητρώα, το ένα το άλλο Ίσως, ε, ναι, να σεβαστούμε, ίσως σεβόμαστε την αρχή της επικορικότητας, αλλά δεν νομίζω ότι, ότι είναι κάτι που είναι εκτός πεδίου και όλα αυτά που λέμε περί σωστής ε, διαχείρισης ε, και ε, για να αποφεύγουμε παρόμοια πράγματα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το καινούριο σαν επιχείρημα, ούτε αλλαγή. Ο κ. Λούντριξον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι σχετικά με τη ε, νομίζω για το 63 θα πρέπει να επιμείνω δεν εντάσσεται στον τομέα αρμοδιοτήτων μας. Τα κάτι μέλη είναι κυρίαρχα από τη στιγμή που πρέπει να ληφθούν παρόμοιες αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, παραμένω σταθερός, επιμένω στο σημείο αυτό. Και διατηρώ τη θέση μου γιατί όπως σας είπα να επαναλάβω και πάλι, δεν είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και αντίθετα φοβάμαι ότι θα μπορούσε να αποδυναμώσει την έκθεσή μας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Θα το δούμε λοιπόν τι θα γίνει ακριβώς. Έχουμε ακόμα μερικές ώρες πριν από την ψηφοφορία και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μπορεί να λάβετε υπόψη σας αυτές τις προτάσεις που σας έχουν γίνει σχετικά με τις συμβαστικές τροπολογίες ε, για να ανασυντάξουμε αυτά τα δύο κείμενα. Θα ψηφίσουμε σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης αύριο Πάμε τώρα στο σημείο 7, το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Γκίρλινγκ. Εξυγχρονισμός πολιτικής δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει το λόγο η συγκήτρια. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ πρέπει να ευχαριστήσω τους και εξηγητέ για το σκληρό του έργο και ακόμη και για τη γραμματεία που μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Διευκόλυναν την εξέβρεση συμβιβαστικών λύσεων. Νομίζω ήταν φτωχή. Μάλλον ήταν καλή. Μάλλον για να βρούμε συμβαστικές λύσει είχαμε περιθώριο, αλλά με μόνον 7 ε, τροπολογίες που αρχικά είχαν ε, υποβληθεί. Δεν είναι ότι δεν θεωρούμε σημαντική τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων και τη δυνατότητά της να προκαλέσει και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την απασχόληση και μάλιστα την ποιότητά της, αλλά περισσότερο υπάρχει πίστη για το πόσο ωφελεί τι μικρότερε επιχειρήσει. Νομίζω αυτό αναγνωρίζεται ευρέω. Κάποιες τροπολογίες ξεφεύγουν λίγο από το πεδίο που κάλυπτε αρχικά η έκθεσή μας, αλλά αυτό νομίζω αστικτοδό το επεδίωξαν κάποια και μίλησαν και για περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία τα είχαμε αναφέρει και νωρίτερα στα πλαίσια των συζητήσεών μας, αλλά νομίζω καλό να το θυμίζουμε ότι και η Επιτροπή ΕΝΒΙ έχει επιληθεί του θέματος αυτού και πολλές από αυτές τις πτυχές στη δική τους νομοθέτηση για αυτή την έκθεση θα επισημανθούν. Κάποια στοιχεία που έχουν προκύψει από τη συζήτηση για τι τροπολογίε είναι η ανάγκη να δημιουργηθούν και άλλε θέσει εργασία, ευκαιρίε. Ξανά και ξανά και ξανά αναφέρεται αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, Πρόεδρε, ποτέ δεν θα πάψει να είναι σημαντικό να περιοριστούν από τη μια ή επαναλήψει και από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι ένα πρωταρχικό στόχο είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερε ευκαιρίε απασχόληση. Κάτι άλλο που αναφέρουν πολλοί οι συνάδελφοι στι τροπολογίε του είναι ότι αυτό το θέμα πρέπει να πλαισιωθεί και να συναρμοστεί με του στόχου τη στρατηγική του 2020. Νομίζω ότι και αυτό το θέμα διατρέχει ολόκληρη την έκθεση. Υπήρξαν βεβαίω κάποιοι τομεί όπου δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Ή δεν βρέθηκε εύκολα συμφωνία, κυρίω. την ε, αντικατάσταση των ε, υπαρχόντων κριτηρίων με κριτήρια ευφύ. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για συγκεκριμένες ιδέες, ε, τις οποίες θα δούμε και με τη μορφή τροπολογιών νομίζω, οπότε θα μπορέσει κανείς να αποφασίσει κάθε φορά ανά την αναπερίπτωση. Συνολικά λοιπόν, ολπίζω ότι θα προχωρήσει το θέμα αυτό στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και μετά την αυρήνη ψηφοφορία ειδικά, ώστε να υπάρχει και η δική μας θέση. Ο κύριος Χιούς και η κυρία Τουρούν. Ο κύριος Χιούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Κέρλινγκ στις εισχογικές της παρατηρήσεις είπε ακριβώς γιατί υπήρξαν προβλήματα με την ε, γνωμοδότηση αυτή. τα ζητήματα που μας μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως και αναφέρονται στις τροπολογίες είναι κυρίως τα από σύμβασης του ΑΕΛΟ του 1994 για τις δημόσιες συμβάσεις το ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ευφύ παρά υπερκριτήρια, το θέμα των υπεργολαβιών και της κοινή ευθύνης. Αυτά είναι ζητήματα που εμείς τα είχαμε για πολύ σημαντικά, αλλά κάπως έχουν ε, παραμεριστεί. Δυστυχώς, ενώ ε, εκπροσωπήθηκα, ε, παρόλο που δεν παρευρέθηκα ο ίδιος στη συνάντηση των σκιωτών για την εξέβρεση συμβαστικών τροπολογιών, πρέπει να εκφράσω δυστυχώς τη λύπη μου που δεν λήφθησαν υπόψη ακριβώς οι δικές μας προτεραιότητες. Στηρίζουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες, ε, την ε κυρίως και όχι τις υπόλοιπες, αλλά εάν υπερψηφιστούν οι τροπολογίες αυτές, θα ζητήσω από τα μέλη της ομάδας μου να καταψηφίσουν όλη την γνωμοδότηση στην τελική ψηφοφορία. Εδώ θέλω να θέσω και ένα ερώτημα στα μέλη του ΕΛΚ σε σχέση με την τροπολογία 40, ε, τροπολογία από μέλος του ΕΛΚ Ζητήθηκε να γίνει ψηφοφορία κατά τμήματα. Νομίζω ότι στόχος είναι να απαλληφθεί δεύτερο τμήμα της τροπολογίας, που αναφέρεται σε θέματα κοινωνικού και δίκαιου εμπορίου, σε θέματα δημόσιων συμβάσεων. Α, τα μέλη του ΕΛΚ να το δουν αυτό ατομικά πιστεύω. Σας ζητώ να σκεφτείτε εάν θα να σκεφτείτε αν μπορείτε να καταψηφίσετε μια τέτοια ε, αναφορά στο κείμενο. Λίγο ακόμα, Πρόεδρε, να ρωτήσω τον κύριο Όρη. Το κατά πόσον λαμβάνει υπόψη τι αλλαγέ που έχουν γίνει στην Ουγγαρία στο δίκαιο περισυμβάσεων, από ό,τι διάβασα θα υπάρξει μείωση και όχι βελτίωση τη διαφάνεια λόγω τη αλλαγή ε, τη νομοθεσία σα. Για δώστε μα μια ιδέα για το τι συμβαίνει εκεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι στο κατάλογο των απορριτών ο κύριο Σωρή, ίσω να θέλει να εγγραφεί τώρα. Η κυρία Τουρούνεν και μετά η κυρία Χίρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στίφεν, θα πρέπει να ξαναδεί τον κατάλογο των ψηφοφοριών, διότι πολλέ από τι δικέ σου τροπολογίε θα ψηφιστούν ούτω ή άλλω πέραν των συμβιβαστικών. Ε, είναι και αυτό μια ιδέα και το βρήκαμε ενδιαφέρον να συμπεριληφθούν. Άρα, ε, περίμενε να δει τι θα γίνει με την ψηφοφορία και μετά κάνει τι συστάσει σου προ τα μέλη τη ομάδα σου. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις τώρα για τα βασικά θέματα της έκθεσης. Εμείς ως πράσινοι έχουμε μια δυσκολία με την τροπολογία 22 των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Το ζήτημα δεν είναι τόσο πολύ πρόθεση πίσω από την τροπολογία, αλλά περισσότερο η διατύπωση. Διότι αυτό που γίνεται είναι ότι ζητάτε η συμπερίληψη των απαρεχόντων υπηρεσίες στι γενικές εξαιρέσεις. Αυτό κατά την άποψή μας είναι κάπως επικίνδυνο και μπορεί να επηρεάσει την αυτοδιαχείριση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Για μας είναι σημαντικό οι παρέχοντες υπηρεσίες να παραμείνουν εκτός του όλου συστήματος της αυτό διαχείρισης. Ίσως να έχετε όμως πιο συγκεκριμένε προθέσεις ε, γι' αυτό που να μην τις έχουμε καταλάβει λόγω διατύπωσης. Εάν βελτιωθεί η διατύπωση, ίσως να συμφωνήσουμε για τις ε, κυρώσεις, τροπολογία 67. Συμφωνώ με την πρόθεση, αλλά θα προτείναμε μια προφορική τροπολογία, διότι ένα κράτο μέλο έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει τι κυρώσει θα επιβάλλει. Αντί να λέμε λοιπόν οι συμβάλλουσε αρχέ είναι υπεύθυνε, θα έπρεπε να λέμε relevant authorities, οι αρμόδιε αρχέ, ώστε να υπάρχει κάποια ευελιξία για το πώ θα επιβάλλονται κυρώσει. Πάντω, η βασική ιδέα να παραμείνει. Ε, προφορική λοιπόν τροπολογία, την οποία την υποβάλλω τώρα μόλι. Και για τι σχέσει δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, μάλλον. Εδώ Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ απόψει. Εγώ πρότεινα να απαλληθεί τελείω η παράγραφο. Ο λόγο είναι ότι, κατά με, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει στο ευρωπαϊκό επίπεδο να εκφράζει προτίμηση για συγκεκριμένε λύσει υπό τη μια την άλλη έννοια. Για να παραμένουμε συνεπεί ω προ τη στάση μα, θα προτείνω την καταψήφιση τη τοπολογία 71 όπου λέγεται ότι οι ιατρικέ σχέσει δημόσιου-ιδιωτικού τομέα δεν αποτελεί καλό εμπορικό μοντέλο. Δεν συμφωνώ. Θα μπορούσε να έχει προστεθέμενη αξία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπαγορεύεται ή να θεωρείται το απόλυτο υπόδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έλεγα λοιπόν να μείνει έξω και να ε, διαγραφεί τελείω η παράγραφο 8. Ολοκληρώνοντα, να πω ότι εδώ η γνωμοδότηση αυτή μάλλον θα είναι χρήσιμη και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ νομίζω θα φανεί αυτό και αν δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας και τις δυνατότητες στρατηγικής χρήσης των δημοσίων συμβάσεων για να ενισχύσουμε και τους κοινωνικούς μας στόχους και στόχους περί απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό θα ε, εμπλουτίσει και την έκθεση της ε, ΙΜΚΟ. Οπότε εμείς ως πράσινοι θα τη στηρίξουμε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χίρς και ο κύριο Κλάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκφράζοντα τον συναδέλφο Κρότσμαν, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Καταρχήν, ο κ. Κρότσμαν ευχαριστεί τη συντάξη σα την γνωμοδότηση για την καλή συνεργασία. Ε, η Άλτε θα υποστηρίξει όλους τους συμβασμούς, ε, τις συμβαστικές τροπολογίες που προτείνονται. Η θέση της ΑΛΤΕ για τις επιμέρους τροπολογίες προσανατολίζονται στις εξής γραμμές. Καταρχήν, οι δημόσιες ε, αρχές θα πρέπει να σέβονται τις ε, κοινωνικές πτυχές στην αρχή της διαφάνειας μη διακρίσεων και αποτελεσματικότητας. Κατά τα άλλα, η χρήση ε, αυτών των δημοσίων αγορών για την επίτευξη κοινωνικής ε, δικαιοσύνης θα πρέπει να, θεωρήσουν, να θεωρηθεί σαν ένα καλό θέμα, αλλά θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Και θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο πεδίο στο οποίο να ωφελούνται και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Εκτός αυτού, όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, νομίζω ότι υπάρχει ήδη κάτι ε, σχετικά και αυτό θα πρέπει να φέρεται και στα εν λόγω έγγραφα. Οι δυνατότητες που υπάρχουν ήδη χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια. Επόμενα σημεία. Η επίλυση του προγράμματος δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την τροποποίηση της οδηγίας όσο από τις πρακτικές κατευθύνες γραμμές. Ε, επαγγελματική ε, μετεκπαίδευση για τις ε, υπεύθυνε υπηρεσίες, ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν σωστά οι ισχύουσες διατάξεις. Στους ορισμένου τομεί όμως ίσως υπάρχει νόημα να διευκολυνθούν οι διατάξεις Ένωση και να καθιστούν πιο ευέλικτες. Θα πρέπει γενικά να γίνονται δεκτές εναλλακτικέ προσφορές για να προωθηθεί η πρωτοβουλία και στον κοινό τομέα. Όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στις ε, ε δημοσίευσεις αυτές ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί ο κ. Κρόσμαν ότι χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Θα πρέπει όμως να αλλάξουν, ε, να εξεταστούν συγγνώμη, εις βάθος ή επιμέρους πτυχές. Η επιτεύξη και πρόθεση εσωτερική αγοράς είναι ένας από τους στόχους των ε, δημοσίων αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα πρέπει για να το πετύχουμε αυτό να ξεπεράσουμε την ε, νομολογία μέχρι τούδε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο κύριος Κρότσμα υποστηρίζει την ε, διαδικασία πρόσβασης ΜΜΕ που πρέπει να βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα, ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάρκ και μετά ο κύριος Άγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην πρώτη παράγραφο της αρχικής πρότασης αναφέρεται ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο στην μόνιμη απασχόληση. Οι δημόσιε υπηρεσίε είναι όμω θέμα τοπική και τοπικών και περιφερειακών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν την ιδιότητα να ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων απασχολήσει σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η υγεία της, απασχόληση απασχόλησης εξαρτάται από την τοπική ή εθνική κατάσταση. Δηλαδή αν το κάποιες εταιρείες τοπικά αυτό θα έχει τοπικούς αντικτύπους. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τη δική μου περιφέρεια της περισμένες εβδομάδες ε, που πρόκειται για τους Bombardier, την ε, επιχείρηση Bombardier που κατασκευάζει ε, σειρμούς και μηχανές και που έχασαν τις, ε, τα συμβάσεις που είχαν στην Siemens. Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις βέβαια στην περιοχή αυτή και στις ΜΜΕ που υποστηρίζουν την Bombardier. Πολλά πρέπει να αλεχθούν λοιπόν όσον αφορά την δυνατότητα του ενίσχυσης από το Ταμείο αντιμετώπιση ε, της ε, Παγκοσμιοποίησης, όπως έχει γίνει με την Ιρλανδία ή με την ε, Αυστρία. Ξέρω όμως ότι οι εργαζόμενοι εκεί στον Τάρβι θα προσπαθήσαν να είχαν διαφορετική υποστήριξη. Ξέρω ότι υπάρχει δυνατότητα μετεκπαίδευσης. Ξέρω αυτοί τι θέλουν. Θέλουν τις θέσεις της εργασία τους. Και δεν τους βοηθάει τίποτα το ότι χάνοντας τη σύμβαση αυτή βλέπουν ότι πηγαίνει σε μια εταιρεία που έχει ε, μια ιστορία διαφθοράς. Τα τελευταία χρόνια η Siemens καταδικάσε σε ένα εκατομμύριο δολάρια από την Γερμανία και την, ε, της ΕΠΑ γιατί προσέφερε κάποια οικονομικά ενάσματα σε εταιρείες που συνεργάζονται. Εκτιμάται παραδείγματο χάρη ότι αυτά που έκανε η Ζήμεν στην Ελλάδα κόστησε στην Ελλάδα δύο δισεκατομμύρια, πράγμα που δεν βοηθάει ούτε την Ελλάδα ούτε εμά. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, ε, αν δεν είναι δυνατόν, η Κομισιόν και το Συμβούλιο να κάνουν ό,τι γίνεται, ότι οι Siemens θα πρέπει να εξεταστεί εις βάθος. Εγώ δεν λέω ότι αυτή η σύμβαση τώρα που πέτυχα την περασμένη εβδομάδα ε, βασίστηκε πραγματικά σε διαφορά, αλλά λόγω του ιστορικού της εταιρεία, εγώ αν σε, μια, ε, σε ένα συμβούλιο για τη δημόσια αυτή σύμβαση, δεν θα έδινα ποτέ τη σύμβαση αυτή στην Siemens. Θα πρέπει να ε, εξεταστεί, γιατί όταν μελετάμε τον εξυγχρονισμό της Πολιτική δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να φροντίσουμε όλα να είναι καθαρά και διαφανή και δίκαια. Ευχαριστώ κύριο Σάντελ και μετά κύριο Παλασά. Σύντομο σχόλιο, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτά που δημιούργησαν στην ΣΥΜΕΣ τα τελευταία χρόνια, ιδίω πρωτοβουλία της NCC, εξετάστηκαν επαρκώς και υπήρχαν πολλές παρεμβάσεις από την πολιτική και τα εποπτικά όργανα για να απογορευτούν και αν υπάρχουν νέες εξελίξεις οπωσδήποτε θα πρέπει να εξαστούν και αυτές. Τώρα για την συγκεκριμένη έκθεση είναι προφανές ότι η προσέγγιση της ηγήτριας διαφέρουν από τις δικές μας, εν μέρη τουλάχιστον. Η συγκέντρια συγκεντρώνεται κυρίως στο θέμα της αγοράς. Εμείς από την άλλη μεριά θέλουμε να δούμε ποια, ποιος είναι ο κοινωνικός προσανατολισμός του μέσου αυτού των δημοσίων συμβάσεων και πώς μπορεί αυτός ο κοινωνικός προσανατολισμός να εισαμοδοθεί. Δεν είναι απαραίτητο ανηφατικά αυτά, μπορούν να συμπληρώσουν τα μέντα δε θεωρώ ότι αυτό που λέει η συγγήτρια ότι κοινωνικά και οικολογικά θέματα δεν έχουν κανένα ρόλο σε μία ε, σύμβαση επειδή εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι ε, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα πραγματικά είναι υπερβολικό μετά η είπε ότι ο κύριος Κρότσμαν, μας διάβασε τουλάχιστον αυτά που τη είπε ο κύριο Κρότσμαν, να μην το πάρετε λοιπόν προσωπικά, αλλά θεωρώ παρόλα αυτά ότι εάν σε αυτή την έκθεση εισαγωγικά αναφέρουμε τον στόχο της έκθεσης αυτής για τις δημόσιες συμβάσεις με, και αιτιολογούμε την δημιουργία διαρκών μέσων απασχόλησης και προστασίας του περιβαλλοντος, θα πρέπει αυτό να είναι και τμήμα των ε, διαγωνισμών για την δημόσια αυτή σύμβαση. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θέμα της πράσινης βίβλου για, τους, ε, για τις και το θέμα των όρων θέσης εργασίας. Τονίζω το ότι απορρίπτεται η σύμπραξη ιδιωτικών και ε, δημοσίων ε, αγορών σύμφωνα με την τροπολογία 70 συγγνώμη, και 71 που θα καταψηφίσουμε. Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε όλες εκείνες τις τροπολογίες οι οποίες κινούνται ιδίω ε, στην κατεύθυνση του, των εφιών ε, λύσεων. γιατί οι ευθύνες λύσεις προωθούν την αηφορία όσον αφορά και την οικονομία και την κοινωνική πτυχή. Προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Έχουμε πολλά αρνητικά παραδείγματα όσον αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις και όσον αφορά ένα dumping μισθολογικό. Και όποιος ε, θέλει να προωθήσει την Ευρώπη του 2020 θα έκανε καλά να τονίσει περισσότερο το θέμα των κοινωνικών συμφερόντων και όχι να αφήνει το θέμα της κοινωνίας και το κοινωνικό εκτός των, της μελέτης αυτής. Ευχαριστώ. Μπαλτασάρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ξεκινήσω απευθύνοντας τη χαρτίριά μου στην εισηγήτρια έδειξε ιδιαίτερη οριμότητα και τέθηκε στη διάθεσή μας με εμπλουτισμό με σημαντικές έννοιες και ακριβώς που χρειαζόταν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ειδικότερα το σημαντικό ρόλο αυτών των δημοσίων συμβάσεων που, έχουν, που μπορούν να έχουν στην όλο θέμα της γενικής ανάπτυξης που χρειάζεται στην Ευρώπη και την ανάγκη όσο γίνεται περισσότερο να απλοποιηθούν οι όλες διαδικασίες, οι όλες προδιαγραφές, έστω και με κριτήρια όμως διαφάνειας και ορθά που να ισχύουν και να είναι κάτι το πιο ευλίγιστο με καλύτερη πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προκήρυξη αυτών των διαγωνισμών που είτε αποκλείονται είτε είναι πολύ περιορισμένη η πρόσβασή τους. Α, λοιπόν, σχετικά με τα θέματα αυτά είναι κάτι το σημαντικό και το θετικό απλοποίηση, μείωση του διαδικαστικού διοικητικού κόστους και ο ρόλος ε, των εταίρων ε, ιδιωτών και δημοσίων. Κάτι που δεν θα πρέπει να αποτελέσει κάτι αρνητικότατο. Θα πρέπει να δούμε στο όλο θέμα που είναι κίνδυνοι, αλλά όχι έτσι πεπαλαιωμένα, ραχνιασμένα να λέμε ότι αυτή είναι ο κίνδυνος της κερδοσκοπία στη σχέση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ίσως ε, απαιτεί ένα τέτοιο κίνδυνο η αγορά. Και κάτι ακόμα, η αλλαγή της διαδικασίας για τη μέγιστη μείωση ακριβώς της ε, προτινόμενης τιμής να ε, είναι κάτι το λειτουργικό και επίσης τα κοινωνικά κριτήρια που θα πρέπει να μπαίνουν στην όλη υπόθεση. Αυτά αποτελούν τις βάσεις ε, που θα μας βοηθήσουν να υπερψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Σημαντικό είναι τώρα να το κάνουμε αυτό και γιατί πρώτοι το κάνουμε και ίσως και η δική μας οι γνώμη να μπορέσει να επηρεάσει τα μέλη της Επιτροπής ΣΥΝΚΟ και επίσης και ε, με τους σοσιαλιστές ε, έχουμε τόση απόσταση που δεν θα είχαμε διαφορετικά δυνατότητα να πετύχουμε κάτι το συγκεκριμένο και τελικό. Και ακόμα σχετικά με τη θέση του ΕΛΚ για την τροπολογία 40. Ζητάμε ξεχωριστή ψηφοφορία γιατί αναφερόμενοι έτσι στα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα. Εμείς συμφωνούμε, αλλά όταν θέλουμε τώρα και άλλα κριτήρια, έτσι, κατά γενικό τρόπο που να έχουν να κάνουν με κάθε τομέα σε αυτές τους δημόσιους διαγωνισμούς, εμείς διαφωνούμε, γιατί κάθε παραμπροκήρυξη, δρόμοι, ε, το ένα τ' άλλο, υπηρεσίες, ε, είναι άλλα τα χαρακτηριστικά και δεν ξέρουμε, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί κάτι τέτοιο, δηλαδή, όχι μόνο να αποδείξει αλλά και να επιβάλλει ε, προδιαγραφές που ορίζει να πάρουμε να δούμε υπόψη μας τον ειδικό χαρακτήρα για την κάθε προκήρυξη. Εντάξει, για τους ασθενήνέστερους είμαστε υπέρ. Όταν έχουμε τώρα γενικά κριτήρια για όλους, τότε το ΕΛΚ διαφωνεί. Δεν είμαστε πεπισμένοι για τον δρόμο που παίρνει πια αυτή η τροπολογία, όπως και άλλες τροπολογίες. Αυτό που ευχόμαστε είναι αύριο να πάμε και να ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Είμαστε έτοιμοι να την υπερψηφίσουμε και σας ευχαριστούμε. Ο κ. Κομφεράτη. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ μεγάλη ευκαιρία, βέβαια λεπτό το θέμα, για να μπορέσουμε να δώσουμε ουσία σε αυτή την αρχή που αναφέρεται στο ξεκίνημα της σύνταξης εδώ ότι ε, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει αποτελεσματικό μέτρο για την πραγματοποίηση της Ευρώπης του 2020. Όχι μόνο σε αυτούς τους δημόσιους προκηρύξεις διαγωνισμών να δοθεί ένα σύγχρονος χαρακτήρας, αλλά να δοθεί και ένα τελικός χαρακτήρας με καταλληλούς στόχους, γιατί υπάρχουν διάφορες απαιτήσει που δεν μπορούν να παρακαμφθούν ούτε να υποτιμηθούν. Πρώτα απ' όλα, ορισμός του πλαισίου των περιορισμών σε αυτούς τις προκηρύξεις ε, και τις προσφορές ε, των εταιριών ε. δεν μπορούμε να έχουμε αποκλειστικά σαν στόχο την μείωση του κόστους, την έκπτωση κάτι το σημαντικό σας στόχο, αλλά δεν επαρκεί για την αποτελεσματικά της εργασίας, προστασία των εργαζομένων και των υπολείπων, αλλά ούτε και παρότριση οικονομική κίνητρο. Θα πρέπει να υπάρξουν και οικονομικοί, κοινωνικοί παράγοντες και στοιχεία και να δούμε και ας πούμε τις προδιαγραφές της πανελλαμβαντικής χώρες αυτά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη βάσει μιας οικονομίας που να μπορεί να συνδυαστεί και να έχει να κάνει και με την πράσινη οικονομία. Εδώ κάνουμε ουσιαστικά ένα έλεγχο, ε, το ανακολουθούμε αυτά που λέμε ότι επιδιώκουμε. Κάτι ακόμα, την όλη αλυσίδα αυτών των αναθέσεων. Ε, από τα πιο επικίνδυνα ήταν ε, ότι η όλη αλυσίδα μεγάλωσε. Ρίχνω μια ματιά σε αυτά μέτρα, στι υπεργολαβίες. Εάν δεν θέσουμε όρια στις υπεργολαβίες, τότε κινδυνεύουμε, επειδή δεν υπάρχει συνοχή, να μην έχουμε αποτελέσματα. Τελευταίο, οι κυρώσει. Πεπισμένος είμαι ότι είναι ε, λάθος ε, να φανταστούμε ότι θα υπάρχουν κυρώσεις εντελώς διαφορετικές η μία από την άλλη. Για ε, να δούμε ας πούμε για τα υπερεθνικά στοιχεία και την απόφαση να έχουμε μια ρύθμιση με κυρώσεις για όσους δεν σέβονται τις συμφωνίες. Και ότι αυτό έχει μια οριζόντια ισχύ με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ε, διαφορετικά θα αφήσουμε έτσι περιθώριο σε άλλα στον τομέα αυτό των ε, προκήρυξεων. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, να είναι όσο γίνεται περισσότερο ομοιόμορφες για να είναι αποτελεσματικές και να μην ε, βοηθούν ε, στο dumping. Η Πρόεδρος. Η συγκήτρια, παρακαλώ, συντομότατη. Έχουμε πολλά σημεία στη μεσιά διάταξη. Εντάξει, η παρέμβασή σας απλό και μόνο είναι ε, για να δούμε αν θα θέλετε να έχουμε αυτά τα νέα αιτήματα. Ναι, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ναι. Είναι αληθέ ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των αγορών και των κοινωνικών πτυχών των ε, ε, δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει να δούμε πού βρίσκεται η ισορροπία. Θα πρέπει να έχουμε κάτι που τελευταία αναλύση είναι ισορροπημένο. Δύο-τρία πράγματα έχω να αναφέρω. Θα ήθελα να παρακαλέσω τα τρια πραγματα έχουμε να αναφερω Δεν ηθελα να παρακαλεσω τα κρατημενα να σκεφτουν τι τροπολογίε αυτέ για τι δημόσιες αγορέ. Εγώ σέβομαι ότι θα μπορούσαν να διαγραφούν γιατί δεν αρμόζουν εδώ. Σκεφτείτε το όμως. Ε, οπωσδήποτε τοποθετείτε γιατί εάν το παραβλέψουμε δεν θα εξαφανιστεί το θέμα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της γνωμοδότησης για να ζήσουμε κάποιες διευκρινήσεις ποιε είναι οι επιπτώσεις των δημοσίων ε, αγορών στις δημόσιες αγορές αυτού του θέματος. Δηλαδή το να γνωρίσουμε, το να γνωρίσουμε, θα ήταν μια πράξη όπως ε, οι στρουθοκάμιλοι που κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο και δεν θα βοηθούσε καθόλου τη γνωμοδότηση. Θα ήθελα επίση να διευκρινίσω ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχουν οι κοινωνικέ πτυχέ στι δημόσιε αγορέ. Προφανώ υπάρχουν. Εγώ αναφέρθηκα σε εκείνα τα θέματα τα οποία είναι μόνο για το περιβάλλον, που δεν έχουν καμία κοινωνική πτυχή. Λοιπόν, σε γενικέ γραμμέ ε, νομίζω ότι συμφωνούμε αρκετά. Έχουμε σαφή κατάλογο ψηφοφορία και θα προχωρήσουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, εγώ σα ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την νομοδότηση αυτή αύριο. Έχουμε ακόμα τρία σημαντικά θέματα στην περσία διάταξη. Σα ζητώ συγγνώμη λοιπόν, αλλά να είστε σύντομοι. Σημείο 8. Ατζέντη για νέε δεξιότητε και θέσει εργασία. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Εξέταση των τροπολογιών τη έκθεση τη κυρία Μπάστο. «455 τροπολογίες υπάρχουν. κυρία Μπαστό, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό καλύπτει πολλά και διάφορα και είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Εδώ έχουμε συστάσεις ε, κλειδιά πραγματικά για τα κράτη-μέλη σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες ε, και για τις νέες θέσεις εργασίες ε, για τα επόμενα δέκα χρόνια πρόκειται για τρομερή πρόκληση. Η πρόκληση αυτή έχει διευκρινιστεί ποια είναι γιατί είχαμε και 365 ε, τροπολογίες όπως είπατε κύριε Πρόεδρε και πρόκειται για πολύτιμη βοήθεια των συναδέλφων. Θα ήθελα άλλωστε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γι' αυτό. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα βέβαια μερικές φορές έχουμε νέες ιδέες, άλλες φορές ενισχύουν προϋπάρχουσες ιδέες και σε ορισμένε έχουμε επαναλήψεις και άλλες δεν συγκεντρώνονται στο βασικό στόχο και ίσως χάνουν την προσανατολισμό των όσων επιδιώκουμε σε αυτήν την έκθεση να σας πω τις ε, μεταβολές που επιφέραμε σχετικά για τις νέες δεξιότητες ε, κλπ. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα περάσματα, μια αναγνώριση επίσης και να καταλάβουμε και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για τα κατάλληλα εκπαιδευτικά όργανα και αρμοδιότητες, δεξιότητες επαγγελματικές ε, που έχουν να κάνουν με τις καινοτομίε, την επιστήμη, την τεχνολογία και για τις υπηρεσίες ας πούμε όπως την υγεία, το άλλο και άλλοι συνάδελφοι ε, νομίζω ότι κάθε ανταπολογίες ενισχύοντας την ιδέα αυτή επίσης η νέα αηφόρος ανάπτυξη στρατηγική του 2020 ακριβώς η κωδικοποίηση των ατόμων που απαιτούν παρόμοια στρατηγική. Και ιδιαίτερα προσέξαμε πρόσεξαν συνάδελφοι ένα θέμα ότι να δούμε ακριβώς ότι απαιτείται μια προσεκτική στρατηγική απέναντι στι πιο βέβαιες ιδέες, ε, γυναίκε παιδιά, άτομα με μειονεκτικά μετανάστες. Επίσης να δούμε την κινητικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιμένουμε πάνω σε αυτό, γιατί δημιουργούν θέσεις απασχόλησης μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις δημιουργούν ανάπτυξη, συνεισφέρουν σε αυτή. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξή τους και καταργώντας τα διοικητικά εμπόδια και δημιουργώντας ένα κατάλληλο πνεύμα συνεργασίας με πολλές παρόμοιες επιχειρήσεις που θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και θα πρέπει να δούμε ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα αναπτύχθηκε είναι η Flexi Security. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάστηκε και αναρωτηθήκαμε πολλά και διάφορα πάνω σε αυτό. Να δούμε πρώτα απ' όλα. Να σας πω ότι εγώ η ίδια ε, ε, Προσπάθησα να ασχοληθώ με τέτοιο τρόπο που να μην τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία. Είπα ακριβώ ότι η security απλά και μόνο ήταν σημαντική και ότι τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προσαρμοθούν στα πλαίσια τα κοινωνικο-οικονομικά. Και είπα ότι δεν, θα, δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος, μια ενιαία συνταγή που θα πρέπει να χρησιμοποιείται παντού σε όλα τα κράτη-μέλη. Με το θέμα αυτό ασχοληθήκαμε αρκετά με αρκετά καλή διάθεση και προσπάθησα να παίξω και εγώ το ρόλο μου σαν εισηγήτρια και θα προσπαθήσω να πετύχω την ε, πιο πλατιά συνένεση πάνω σε αυτό ώστε αυτή η σημαντική πτυχή να μας βρει διηρημένους αλλά, αλλά μόνο να μας συνενώσει και να μας βοηθήσει να υπάρξει μια σχετική κατάλληλη διευκρίνηση σε αυτήν την έκθεση. Ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ ευαίσθητο για κάποιες πολιτικές ομάδες και ιδίως ό,τι αφορά το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στα διάφορα κράτη-μέλη και εδώ στις τροπολογίες ε, φάνηκε αυτή η ευαισθησία. Αυτό που πρέπει ήδη να πω είναι ότι μελετούμε με πολύ προσοχή όλες τις τροπολογίες και τις 85 και βρισκόμαστε στη φάση εξέβρεση συμβαστικών λύσεων. Ήδη 34 έχουν ετοιμαστεί. Για τις τροπολογίες που μπορούν να γίνουν αποδεκτές και επικεντρώνονται στα βασικότερα μηνύματα που πρέπει να περάσουν ε, με την έκθεση αυτή. Και επίσης περιμένουμε και το αποτέλεσμα των γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Γυναικών και της ΣΥΤΡΕ, προκειμένου να εγκριθούν και τις ε, επιτροπές αυτές και από το Σεπτέμβριο πια σε συνεργασία με τους κοιόδους συζητητές να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε μία σύνταξη πλέον της έκθεσης καλύπτοντας και τις τροπολογίες που θα έχουμε εντωμεταξύ μεταξύ επεξεργαστεί ώστε οι συνάδελφοι να έχουν και περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους για να σκεφτούν. Ευχαριστούμε η κυρία Πλόμ και η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Ως σκιώδης εισηγήτρια της ε, ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, να πω ότι έχω αποβάλει 70 τροπολογίες από τις 300 τόσες. Νομίζω ότι πραγματικά προσπάθησα να επικεντρωθώ σε στατηγικές πτυχές της έκθεσης αυτής. Έκθεση που επιμένει στην ανάγκη υιοθέτηση μια σειρά ιεραρχημένων στόχων. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι σε ό,τι αφορά την ευκαιρία να αναλυφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να καλύψουμε τις ανάγκες των πλέον ευάλωτων, νομίζω ότι αυτή η μερίμνα είναι σημαντική. Ίσες ευκαιρίες πρέπει να υπάρχουν για όλους ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ε, Επιτέμφαση έμφαση δίνεται μέσω των τροπολογιών στην ασφάλεια. ένα εργαλείο σημαντικό για την ε, εκπαίδευση των εργαζομένων και τη διαρκή τους ενημέρωση. Πρέπει να προστατεύονται οι εργαζόμενοι ως προς τα κοινωνικά τους δικαιώματα και ε, έναντι της ε, ανεργίας. Επίσης, οι διαχωρισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασία είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εξέφρασα και την ικανοποίησή μου για τη δράση τη εκτελεστική επιτροπή, ως προς την αναζήτηση εργασίας. Πιστεύουμε ότι όντως κάθε εργαζόμενος, κάθε κατους μέλου πρέπει να καλύπτεται από νομικές εγγύσει. Ιδίω ω προς την καταπώνηση τη οποία μπορεί να πέσει θέμα. σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί αυτό, δεν είναι δυνατόν να συμβαστούν ο οικογενειακός με τον επαγγελματικό βίο και να προστατευτεί και η υγεία του ίδια. Επίσης, καταδικάζεται η διακριτική μεταχείριση που ήδη βλέπουμε να πλήττει πολλές φορές τους λάθρομετανάστες και βεβαίως οι διακρίσεις ε, με βάση το φύλλο δεν θέλουμε να εξακολουθήσουν στην ε, αγορά εργασία. Η κοινωνική οικονομία, η social economy όπω την ονομάσαμε, θα μπορούσε να, να γίνει ένας χώρος για δημιουργία περαιτέρω θέσεων απασχόλησης. Επίσης αναφέρθηκα στην απόσπαση εργαζομένων, κάτι που αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στην περίοδο κρίσης και θα χρειαστεί νομική ρύθμιση. Και μετά αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το υπενέχθηκα και προηγουμένω. Αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί στι επενδύσει. Παραγωγικέ επενδύσει, λαμβάνοντα υπόψη τι πραγματικότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι διαφορετικέ. Υπάρχουν νέε αρμοδιότητε ω προ την βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν, οφείλουν να προωθήσουν τις οικολογικές μέρημνες προκειμένου να αντιμετωπιστούν και τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να διευκολυνθεί και η μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές σε άνθρακα Πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να σκεφτεί πώς θα εισαχθούν νέες καθοριστικές αρμοδιότητες που να αφορούν το περιβάλλον, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, και την βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον αναφέρομαι στις τροπολογίες μου και στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των νέων της αρμοδιοτήτων και το πώς όλα αυτά μπορεί να συνεισφέρουν στην τόνωση της απασχόλησης. Νομίζω ότι με τους υπόλοιπους και όδης εισηγητές και σε συνεργασία με την εισηγήτρια Μπαστός μπορούμε να καθορίσουμε σωστά την στάση του Κοινοβουλίου εδώ σε ένα τόσο σημαντικό τομέα. Κύριε Χάρκιν, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Και επειδή βρισκόμαστε προ το τέλο τη ημέρα διάταξη, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά διαθρωμένη και σφαιρική η έκθεσή τη. Αυτό δεν ξέρω τι θα πρέπει να μα πει για τι 365 τροπολογίε, αλλά πραγματικά σα εύχομαι καλό κουράγιο. Και να βρείτε και συμβαστικέ λύσει πολύ σύντομα. Κάποιε από τι τροπολογίε που εγώ προτείνω ασχολούνται με θέματα όπω η πρόσβαση στην οικονομική στήριξη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, την κοινωνική οικονομία που αναφέρει και συνάδελφο, την προώθηση ενό ποιοτικού πλαισίου για, τα, για τι μαθητείε, για την εκπαιδευτική έργαση, τι ασκήσει μάλλον, για την άτυπη μάλιστα εκπαίδευση, να μην ξεχνάμε και τον εθελοντισμό, ε, ε, ευρωπαϊκό έτο εθελοντισμού φέτο. Ελπίζω ότι θα τις στηρίξετε τις περισσότερες, καθώς πολλές ήδη απηχούνται στις συμβαστικές σας λύσεις. Κάτι άλλο που βρήκα ενδιαφέρον, το ανέφεραν και κάποιοι από τους συναδελφούς, να δούμε τους βασικούς τομείς που εδώ αναφέρονται, πράσινες εργασίες, επίσης πολύ σωστά ο τομέας παραγωγής τροφίμων της Γεωργίας. Είναι και αυτό κάτι που θα μπορούσε να απασχολήσει την ε, Επιτροπή μας. Επίσης, πολύ ανέφεραν το θέμα των φίλων. Και κάποιοι ανέφεραν, όπω η κυρία Χάρκιν, τη διαβίου κατάρτιση και την εκπαίδευση. Και αυτό καλό θα ήταν να καλύπτεται από τι συμβαστικέ σα λύσει. Η κυρία Σφέτερ. Ja, vielen Dank. Ich kann es sehr kurz machen, weil meine Vorrednerin äh, schon wesentliche Punkte. Ε, θα είμαι σύντομη γιατί η προλήψη σα ανέφερε διάφορα θέματα που μπορώ να υποστηρίξω και είναι πολύ καλό να καταλήξουμε σε κοινέ καλέ ε, τροπολογίε και θα θέλουμε σύντομα να μάθουμε ποια μορφή έχουν οι συμβαστικέ ε, λύσει. Ε, να έρθετε σε επαφή σα μαζί μα το γλυγορότερο δυνατόν λοιπόν για αυτά. Καλό θα ήταν. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία τη Κομισιόν ε, για τι νέε δεξιότητε και νέε θέσει απασχόληση ε, σχετίζεται και μία πρωτοβουλία για νέε θέσει απασχόληση. μόνο ε, και λήφθη υπόψη μια τροπολογία επανερχόμενη στην, στο κίνημα που είχε ήδη ε, υιοθετήσει το Κοινοβούλιο και όπου εξαιρέθη εκείνος ο τομέας ο οποίος αφορά άμεσα την πρωτοβουλία της Κομισιόν για τις νέες δεξιότητες. Θα ήταν πολύ καλό να διατυπώσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και τις συμβαστικές τροπολογίες σας. Ένα δεύτερο θέμα που έθιξε και πάλι η κυρία Πλάμ είναι ότι θα πρέπει να φροντίσουμε αυτές οι νέες δεξιότητες για νέες θέσεις απασχόλησης δεν είναι μόνο στο επίπεδο υψηλών δεξιοτήτων, αλλά σε όλους τους τομείς. Και θα πρέπει να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εκείνους που έχουν λίγες δεξιότητες, που είναι άσχημα εκπαιδευμένοι, δηλαδή δεν είναι πολύ εκπαιδευμένοι. Και εκεί θα πρέπει να συγκεντρώσουμε κυρίως την προσοχή μας. Ξέρουμε επίσης ότι ιδίω για την αηφόρα οικονομία, εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο δυναμικό θέσεων απασχόληση και γι' αυτό θα θέλουμε να συγκεντρώσουμε το προσοχή σε αυτή την ομάδα. Αυτά είναι τα ε, κεντρικά στοιχεία που έχουμε στι τροπολογίε και θα ήταν πάρα πολύ καλό η συγγήτρια να λάβει υπόψη αυτά τα σημεία όσον αφορά το περιεχόμενό του και να το τονίσει στι δικέ συμβαστικέ προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Μαστός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπαν οι συνάδελφοι που υπέβαλαν τροπολογίες κάτι που και εγώ προσπάθησα να το πω προηγουμένως. Μιλάμε για ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και ευρύτατες συζητήσεις για θέματα που ήδη τα έχουν καλύψει με ανακοινώσει τη Επιτροπή, όπω η απασχόληση ή άλλα που μα απασχόλησαν και στη σημερινή διάταξη σήμερα. Μετά την οικονομική κρίση και την κοινωνική κρίση, τι συνέπειέ τη που ακόμη ζούμε. Κάτι που όλοι οι συνάδελφοι ανέφεραν και τις ευχαριστώ όλες για τις παρεμβάσεις τους και τις τροπολογίες που υπέβαλαν. Πρώτα απ' όλα, η καταπολέμηση, μάλλον η στήριξη της οικονομίας της Ευρώπης ε, και του κάθε κατου μέλους, ώστε τώρα στο μέλλον το έγγραφο δεφό που ετοιμάστηκε ως ακρογωνιαίος, δεν θα κουράζομαι το επαναλαμβάνω, λίθος, για το πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα εργατικά μας συστήματα, τις οικονομίες της Ευρώπης και με τις ε, ανησυχίες που ανέφερε το έγγραφο της Επιτροπής και τις μέρες που δεν εκφράστηκαν μέσα από την συζήτηση. Το θέμα είναι τεράστιο, είναι ευρύτατο και βλέπω να απασχολεί τους πάντες. Από τις τροπολογίες λοιπόν η βασική ανησυχία που προκύπτει με οθεί να αναζητήσω μια κατάλληλη συμβιβαστική λύση, μια, με τη σωστή διατύπωση και θα συνεργαστώ στενά γι' αυτό με τους Σκιώδης εισηγητή. Δεν έχουμε πάρα πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα. 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή το θέμα αυτό, ήδη την προσεχή εβδομάδα. Πολλοί συνάδελφοι θα έχουν φύγει στα κράτη-μέλη τους, στις εκλογικές τους περιφέρειες ή στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου Οπότε, κάτι που ούτως ή θα το θυμίσω στους συναδέλφους με mail, στις 6 Σεπτεμβρίου θα βρεθούμε με τους σκιώδεις εισηγητές, το λέω και εδώ, για να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις συμβαστικές λύσεις που θα έχουν προταθεί. Ως τότε, προσκαλώ όλους όσους ενδιαφέρονται να μας δώσουν ιδέες για συμβαστικές λύσεις, ώστε το Σεπτέμβριο να ξέρουμε τι θα συζητήσουμε. Και να είναι και λίγο πιο αποσαφηνισμένη η ημερήσια διαταξή μας για να δούμε τι θα κάνουμε με όλες αυτές τις τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο για τη σύνταξη των συμβαστικών προτάσεων. Σας έχουμε όμως εμπιστοσύνη. Κατόπιν αιτήματος της ηγητού μας φτάνουμε στο σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης ζήτημα τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Κυρία Εισηγητριά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ που το εξετάσετε τώρα αυτό το σημείο. Η πρόταση είναι να ε, προϊοθετήσουμε αυτή την έκθεση με την απλουστευμένη διαδικασία και χωρίς τροπολογίες. Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτός ο κανονισμός σας σαν στόχο να παρατείνει το κοινωνικό ταμείο μέχρι το 31 Δεκεμβρίου 2013. Δηλαδή 18 μήνες ε, και αν αφαιρέσουμε και στερινές διακοπές 15 ε, μήνες, 16. Πολύ σύντομη χρονική περίοδος και εάν υποβάλουμε τροπολογίες δεν θα προλάβουμε νομίζω να τις συμφωνήσουμε πάνω σε αυτές έγκαιρα. Η Κομισιόν επίσης θα υποβάλει κάποιες προτάσεις φέτος στο φθινόπωρο για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης μετά το 2013 και τότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να προτείνουμε κάποιε ε, σημαντικές αλλαγές. Προτείνω λοιπόν να έχουμε ένα ψήφισμα από την τροπή Απασχόλησης για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις δικές μας απόψεις. Τέλος, έχω να πω ότι αυτός ο κανονισμός που παρατείνει την περίοδο εφαρμογής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 διατηρεί το ποσοστό χρηματοδότηση στο 65%. Δύο γενικά σχόλια. Καταρχήν, οι λόγοι για την παράταση. Σύμφωνα με την άποψη τη Κομισιόν, τα ποσοστά ε, ανεργίας είναι στα γύρω τα 9% για το 2011 και 2012 προβλέπεται να μείνουν εκεί γύρω στους 9 και κάτι λίγο. Σε ορισμένα κρατημέλη βέβαια είναι πιο ψηλά από ό,τι σε άλλα χρόνια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο ανεργίας είναι πάρα πολύ υψηλό. Και γι' αυτό το κοινωνικό δεν θα πρέπει να απορροφήσει κάποια του προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Επίσης η Κομισιόν λέει ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών που απάντησαν στις ε, διαβουλεύσεις αυτές θεώρησαν ότι είναι καλή αυτή η παράταση. Αλλά βέβαια δεν ξέρουμε πόσα κράτη ανταποκρίθηκαν. Το ότι εκείνα που ανταποκρίθηκαν συμφωνούσαν δεν μας λέει πολλά. Λοιπόν, δεν ξέραμε αν ήταν μια πλειοψηφία, μια μεγάλη πλειοψηφία, καθόλου πλειοψηφία. Εξετάζοντας τον προπολογισμό του 2012 και τις περικοπές για το Συμβούλιο, επίσης δεν πήραμε κάποιες πληροφορίες από την Πολωνική Προεδρία σήμερα για το τι έχει κατά νου το Συμβούλιο για το Ταμείο αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή καμία ένδειξη. Τέλος. Εξετάζοντας τώρα τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη, το ξέρουν αυτό, το Ταμείο δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει τα 500 εκατομμυρία σε ένα τρέχον έτος. Το 2010 το ποσό που ζητήθηκε ήταν 132 εκατομμύρια και το 131 και προηγουμένως ήταν πολύ λιγότερο. Λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Παρόλο που αυξάνονται τα ζητούμενα ποσά, παρόλα αυτά ε, πόρο απέχουν από το ανώτατο όριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, ξέρω των σοσιαλιστών να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για τον τρόπο προσέγγισής σας ε, και ότι συμμερίζομαι τις προτάσεις σας ε, στην Ολομέλεια να επωφεληθούμε από τη συζήτηση και για να συμφωνήσουμε στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ανανέωση αυτού του μηχανισμού που λέγεται μηχανισμός κρίσης και να υποφεληθούμε από αυτές τις ευκαιρίες μέσω ενός ψηφίσματος παρουσία του Επιτρόπου για να ασχοληθούμε με διάφορα σημεία σημεία που μας απασχολούν για τη συνέχεια. Πάνω συμμερίζουμε την ισχύ σας για τη φύση της όλης συζήτησης στο Συμβούλιο. Το είδαμε ήδη στην συζήτηση με την Πολωνική Προεδρία. Κάπως ε, ταρακούν, συνήθηκαν τα πράγματα ίσως και δεν ξέρω αν θα μπορούμε να είμαστε ακριβώς ενήμεροι των ε, τοποθετήσεων των διαφορών κρατών μελών ε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Τώρα για το θέμα το πώς αυτός ο μηχανισμός θα επεκταθεί και στη γεωργία αυτή η ανάληψη υποχρέωσης για τη μείωση του προβλήματος της ΚΑΠ πώς να το πούμε Εντάξει, όλες οι υπόλοιπες πολιτικές θα πρέπει να απορροφήσουν μέρη της ΚΑΠ. Το είδαμε ακριβώς για την τραπεζα τροφίμων και τώρα για το αρμόδιο σχετικά με την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει να δούμε τις οικονομικές πολιτικές ε, και όλες θα λάβουν ένα αγροτικό χαρακτήρα. Προσπαθώ να το πω, αλλά αυτό θέλω να πω. Να βάλουμε και ψήγματα αγροτικής, ε, αγροτικών πτυχών εκεί. Εντάξει, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στον τομέα αυτό. Από τη στιγμή που επιθυμούμε αυτός ο μηχανισμός να επεκταθεί και σε διάφορες πτυχές αγροτικές, έχουμε μπροστά μας μια διάσταση και της παγκοσμιοποίησης και το τι γίνεται με την κρίση που ίσως, ίσως μας οδηγήσουν και σε υποβολή αντιπροτάσεων και στην όλη λειτουργία του ε, Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση να συμπεριλάβουμε και διάφορα στοιχεία αναδιάρθρωση όπως ακριβώς εδώ και εκεί έχουμε συναντήσει και που είναι στα πλαίσια όλου αυτού του εργαλείου να δούμε όμω και τι μπορούμε να αναφέρουμε στην πρόταση ψηφίσματο που ελπίζω παράλληλα να μπορέσουμε να ψηφίσουμε με την επαναφορά ακριβώ του μηχανισμού κρίσης, ελπίζοντας ότι θα συμβούν τα πράγματα και θα υιοθετηθούν με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο. Η Επιτροπή είναι παρούσα από ό,τι γνωρίζω. Μισό λεπτό πριν λάβει την λόγο κάποιος από την Επιτροπή, κάποιος άλλος από εσά, ο κ. Μπουλάν. Όχι εσείς, κυρία μου, όχι. Γραμμάς Επιτροπής, ε, μήπως θα θέλετε να λάβετε το λόγο. Ούτε εσείς. πολύ καλά. Υπέροχα. Κύριε Χάρκιν, θέλετε και εσείς να λάβετε το λόγο. Ούτε εσείς. Ε, εντάξει, εντάξει. Εσείς ναι. Ε, Όχι. Ούτε εσείς. Μη μου φεύγετε, μη μου φεύγετε. Θα πρέπει να κάνω τις ανακοινώσεις μου. Με τον τρόπο αυτό όμως προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Πώς, όχι μη. Καμία τροπολογία. Τι κάνουμε. Παλαβάνω. Θα ψηφίσουμε Λοιπόν, κύριε εισηγήτρια, κύριε, η εισηγήτρια θα μας προτείνει, θα μας υποβάλει μια πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με αυτά της Επιτροπής και εμείς θα αποφανθούμε σχετικά. Έτσι, παίρνουμε την κατάλληλη πορεία για να έρθουμε λοιπόν τώρα στις ανακοινώσεις. Να σας πω ότι έχουμε έτοιμα για δικαίωμα διαμονής και εργασίας μετά από τις 22 Ιουνίου, τον τριμερή διάλογο, πετύχαμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή μας ε, να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία. Μετά δε από αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθη με το Συμβούλιο, που έκλεισε με το Συμβούλιο, οι δύο επιτροπές είπαν και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά θετικό με κατάλληλη συνεργασία χάρη σε, μεγάλο μέρος της όθησης ε, του συγγητού μας και η Επιτροπή Λιμπέ θα πρέπει να απευθύνει στους αντιπροσώπους του Κορεπέρ ένα μήνυμα για το τρόπο της διαδικασίας συναπόφασης και να εκφράσουμε την σύμφωνη γνώμη μας τώρα συγητής, μήπως θα επιθυμούσα το λόγο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την ερμηνεία σας, κυρία Πρόεδρε. Μόνο μια παρατήρηση. Αυτά τα δύο σημαντικότερα που ζητάει η Επιτροπή μας έγιναν σεβαστά από την Επιτροπή, από το Συμβούλιο, από την Επιτροπή Λίμπε αλλά όχι μετά από δικές μου προσπάθειες, αλλά από τις προσπάθειες της Προέδρου της Επιτροπής. Συνάδελφε, η συλλογική ενέργεια και ξυπνάδα μπήκε στη μέση και λειτουργήσε και χαίρομαι γι' αυτά. Λοιπόν, έχετε αρκετές συνεκκοινώσεις, μη σας θα τις πω τώρα αριθμητικά, αλλά σας προτείνω να υιοθετήσουμε τα πρακτικά της 20 της 4ης 25 Μαΐου, 6ης Ιουνίου, 15-16 Ιουνίου να εγκριθούν τα πρακτικά. Εντάξει, καμία παρατήρηση άλλη. Τα πρακτικά λοιπόν αυτά εγκρίνονται. Σας ευχαριστώ. Σεβαστήκαμε και το ωράριό μας. Αύριο στις 9 το πρωί παρακαλώ τις καρτούλες για να ψηφίσουμε, έτσι.